Bien, Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε ημερήσια διάταξη φορτωμένη. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει για τα πρακτικά τη προηγούμενη συνεδριάσεω του, το συνεδριάσεω του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, θεωρούνται συγκεκριμένα τα πρακτικά και θα ήθελα να γίνει ανταλλαγή απόψεων αυτή που προβλέπετε όσον αφορά την επόμενη έκθεση της Υποεπιτροπής έκθεση που ασχολείται με τεχνολογική βιομηχανική βάση της αμυντικής ε, βιομηχανίας Ευρώπης ο Μάικλ Γκάλερ ε, θα είναι εισηγητής είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής στο τέλος του έτους είναι στη μέση διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Προβλέπονται συζητήσει. Τρει πτυχέ τη άμυνα Ευρώπη. Ένα, ποια είναι η ορατότητα τη πολιτική ασφαλεία και τη άμυνα. Άλλη πτυχή, οι όλε τι δυνατότητε που υπάρχουν. Και τρίτη πτυχή είναι η αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη. Άρα θα ήταν σκόπιμο γρήγορα, με τον αξιωτικότερο τρόπο που γίνεται, με του συναδέλφου τη ΣΥΤΡΑ, να συντάξουμε μια έκθεση επί της ουσίας των ζητημάτων που είναι αποφασιστικής σημασίας. Μάικλ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ε, ξέρετε, ε, προετοιμάζουμε ε, αυτή τη στιγμή πυρετοδός ε, της, ε, της συνεδρίαση του Δεκεμβρίου που θα είναι αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για θέματα αμυντικά και περιμένουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αύριο θα συνέλθουν τα Υπουργεία Οικονομικών, τα Υπουργεία ε, άμυνας για να τοποθετηθούν στην ανακοίνωση της Κομισιόν και εντωμεταξύ περιμένουμε και την ανακοίνωση της κυρίας Άστον. Κατά διάρκεια λοιπόν των ε, διαπραγματεύσεων νομίζω ότι υπάρχει και ρόλος για το κοινοβούλιο μας, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η φωνή των 500 εκατομμυρίων θα ακούγεται και στην ε, άμυνα, στην ΚΕΠΑ. Η αμυντική βάση είναι πολύ σημαντική και αυτό δεν πρέπει να είναι στα χέρια μόνο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Είμαι επίσης πεπισμένος ότι με τις δραστηριότητές μας ε, θα κατορθώσουμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε στη συνάντηση κορυφής ε, να, από αυτή να προκύψουν ε, καινούργια ρεθίσματα. Εγώ θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια λειτουργική, αποτελεσματική κοινή αμυντική πολιτική και χρειαζόμαστε και την δική μας την ευρωπαϊκή ε, βάση εξοπλισμών. Και θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι αυτός σκοπός. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι στο πλαίσιο αυτής της ευρωπαϊκής αμυντικής ε, πολιτικής ε, θα πρέπει να βρεθούν εξοπλισμοί που θα είναι οικονομικοί και που θα μπορούν να παραδίδονται την κατάλληλη χρονική στιγμή έτσι ώστε να μπορεί κανείς να ανταποκριθεί ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η βάση των εξοπλισμών θα πρέπει να είναι οι απαιτήσει που ήδη έχουν εκφραστεί για να επιτύχουμε το στόχο μας. Η σημασία του θέματος μας είναι γνωστή εδώ και πολύ καιρό. Σας ε, παραπέμπω ε, σε αυτά που έχουν πει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Άμυνας, τα Υπουργεία Άμυνας της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά ήδη από τον Ιούλιο του 2000 στο πλαίσιο που αφορούσε την αναδιάρθρωση της ε, ε, το τομέα εξοπλισμών. Ε, Επίσης ε, υπάρχει μια στρατηγική που αφορά στην ενίσχυση ε, της ε, πολιτικής των εξοπλισμών και στην στρατηγική ETIP, η οποία εγκρίθηκε το 2007. Διερωτώ με βέβαια ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της πολυμερούς ευρωπαϊκής στρατηγικής και διερωτώ με γιατί για την Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει ε, εκτέσεις ε, εφαρμογής. Επάνω σε αυτά θα βασιστεί η έκθεσή μου και σε τελική ανάλυση, κατά την άποψή μου, το κοινό μας καθήκον είναι να αναφέρουμε ε, πού μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τη μέχρι τώρα εφαρμογή και πού είναι απαραίτητο να γίνουν και άλλα βήματα. Επίσης υπάρχει απόλυτη συμφωνία ότι όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες τόσο στον τομέα της ζήτησης όσο και της ε, προσφοράς. Και θέλω καταρχήν να μιλήσω για τη ζήτηση, δηλαδή πώς είναι δυνατόν τα 27, σύντομα 28 κράτη να ε, περικόπτουν τους ε, προπολογισμού άμυνας χωρίς συντονισμό και χωρίς να προσπαθούν να καθορίσουν κοινή ευρωπαϊκή πράξη. Για μένα είναι λογικό πρώτα απ' όλα να καταστήσουμε σαφές τι διαθέτουμε, τις ε, δυνατότητες των κρατών μελών. Αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν σε έναν ευρωπαϊκό απολογισμό. Και πάνω σε αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε τι ακριβώς χρειαζόμαστε για να ξέρουμε και τι μπορούμε. Οι απαντήσεις αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια ευρωπαϊκή λευκή βίβλο έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τη ζήτηση. Για να υπάρξει ε, πραγματικά μια διαδικασία ευρωπαϊκής εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής θέματα. Εναρμόνιση των απαιτήσεων, σύνθεση της ε, ζήτησης και συντονισμός ε, της ε, παροχής και στο τέλος συντονισμένη χρήση και βελτίωση των συστημάτων. Τα παλαιότερα παραδείγματα όπως το A4M ή το Tiger, τα συστήματα αυτά εξοπλισμού δείχνουν ότι υπάρχουν πολύ καλές ε, προθέσεις, όμως ε, αυτές οι προθέσεις τελικά υπονομεύτηκαν λόγω ειδικών εθνικών συμφερόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στον τομέα της ε, τυποποίησης και των προδιαγραφών. Ας πούμε, το software defined radio, το software των ασυρμάτων όπου πέρα από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές μπορούμε να ορίσουμε και τις παγκόσμιες προδιαγραφές. Επειδή έχουν χαθεί χρήματα και χρόνος λόγω του ότι υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στις εθνικές προδιαγραφές και υπάρχουν και διαφορετικά συστήματα πιστοποίησης, αυτό που παίζει ρόλο είναι τα κράτη-μέλη και οι οργανισμοί πιστοποίησης και η Επιτροπή να βρουν κάποια λύση έτσι ώστε να διευκολύνουν τη διασυνοριακή πιστοποίηση και να διαμορφώσουν τη μακροπρόθεσμη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Υπάρχει αυτή η σκέψη και υπάρχει και η σκέψη που αφορά το στάνακ του ΝΑΤΟ και διαρωτώ με πού ήταν οι προδιαγραφές του ΝΑΤΟ όταν ε, η ε, Επρόκειτο να στηριχθούν τα γαλλικά τζετ στο Μάλι από τους Γερμανούς με ένα αέριο ανεφοδιασμό. Ε, τότε όμως αυτό δεν ήταν δυνατόν γιατί οι αντλίες δεν ήταν συμβατές. Εγώ λοιπόν ε, θεωρώ ότι οι προδιαγραφές του ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ ευρείες. Η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι πολύ ανώτερη από το σύστημα ΣΤΑΝΑΚ οι ε, στρατιωτικές επεμβάσεις στο Αφγανιστά και στη Λιβύη κατέδειξαν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει security of supply, ασφάλεια στον ε, ανεφοδιασμό ή στον εφοδιασμό. Και ε, εδώ πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο πλαίσιο τα ευρωπαϊκά κράτη ε, έχουν συνεργασία σε θέματα νομισματικά, αλλά αυτή η εμπιστοσύνη δεν υπάρχει στα αμυντικά. Αρκεί να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν μεμονωμένες ε, περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να γίνονται και εξαγωγές μέσα στην την Ευρωπαϊκή Ένωση εξοπλισμών. Αυτό όμως είναι απαράδεκτο, γιατί με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού. Ε, τα κράτη-μέλη γιατί δεν μπορούν να δίνουν αμοιβές ε, υποχρεώσεις ε, για γενικές ε, εγγύσεις εξαγωγών. Ίσως το βήμα αυτό θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης ή συνεργασία μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του Eurogroup ή του Schengen. Βέβαια εκεί υπάρχει μια πραγματικότητα, μπορεί να επεκταθεί και περαιτέρω. Η έκθεσή μου εστιάζεται σε σημαντικές ε, τεχνολογίες, Key Enabling Technologies. Υπάρχει ανακοίνωση της ε, Κομισιόν, μια ευρωπαϊκή στρατηγική ε, για τέτοιου είδου ε, τεχνολογίε θα μπορούσε να δημιουργήσει θέσει εργασία. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Ιουνίου του 2012. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο το θέμα αυτό να επεκταθεί και σε τομεί ε, ασφάλεια και άμυνα. Ο στόχο είναι η Κομισιόν να αναλάβει την εντολή να προσφέρει απεριόριστη προσβασιμότητα, μάλλον το ξαναλέω ο στόχος είναι να δοθεί εντολή στην Κομισιόν να καθορίσει μια στρατηγική για απεριόριστη διαθεσιμότητα τεχνολογιών οι οποίες είναι καθοριστική σημασίας για την άμυνα και την ασφάλεια. Υπάρχει η σύσταση για την τεχνολογία του διαστήματος και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προσφέρουμε και ε, την τεχνολογία στην άμυνα μέσα από την μικροτεχνολογία και την νανοτεχνολογία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορα προγράμματα πλαίσιο και κατόπιν τούτου διαθέσει ειδική τεχνογνωσία. Πρέπει λοιπόν να διασφανιστεί ότι η συμβαστική λύση για την έρευνα ε, πρέπει να οδηγεί σε συγκεκριμένη εφαρμογή. Όσον αφορά το μέλλον, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δω ε, τι ακριβώς ε, θα προτείνουν οι προτάσεις της Επιτροπής για την έρευνα στην άμυνα στην Ευρώπη. Χαιρετίζω την πρόταση που έχει κατατεθεί και εύχομαι με βάση αυτά τα προκατρακτικά μέτρα να ε, ενισχυθεί η έρευνα και να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2009 ενέκριναν το αποκαλούμενο αμυντικό πακέτο, τότε κατέστη δυνατόν να επεκταθεί η κοινή αγορά και στα εξοπλιστικά. Υπήρχαν ε, βέβαια κάποιες ε, επιφυλάξεις ε, στο πλαίσιο του άρθρου 346. Αυτές δικαιολογούνται από το άρθρο αυτό, πρέπει όμως να αιτιολογηθούν. Τώρα αυτό που παίζει ρόλο είναι οι κρατικοί οργανισμοί προμηθειών τις ευρωπαϊκές, τους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς να τους παγιώσουν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει γραφειοκρατία και αυτή όμως δεν πρέπει να θέσει κίνδυνο την επιτυχία της ευρωπαϊκής κοινή αγοράς. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα τα οποία προτείνω και έτσι λοιπόν αν μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά νομίζω ότι θα διαμορφώσουμε ένα πολύ καλό πλαίσιο για την διασφάλιση της εξοπλιστικής βάσης στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις ε, πολιτικές αγοράς και εκτός Ευρώπης διότι η ε, διαλειτουργικότητα ε, δεν εξυπηρετείται με μεμονωμένες αγορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μίκαελ για αυτές τις πρώτες σαφείς και πολύτιμες ε, αναφορές σου. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για το θέμα σήμερα και δεν έχουμε και έγγραφα που να έχουν διανεμηθεί θα ήθελα η συζήτηση να γίνει αρκετά γρήγορα. Θα ζητήσω τον Ζαν Πιέροντι, που εκπροσωπεί την Επιτροπή Ήτρε, να πει μερικά πράγματα, αν θέλει να προσθέσει κάτι. Και μετά έχουμε τον κ. και την κυρία Λέζινγκ, που είναι σκιώδεις εισηγητές και επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Ο Ζαν Πιέρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, εν ονόμα της Επιτροπής Βιομηχανίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη δική σας επιτροπή που απεδέχθη την αρχή του άρθρου 50 για την συνεργασία των, των επιτροπών μας και έχω επιφορτιστεί στη συνεργασία με τον κύριο Γκάλερ που γνωρίζω πολύ καλά και είναι μέλος ε, πολύ ποιοτικό να κάνω τα αναγκαία στα πλαίσια της συνεργίας των αρμοδιοτήτων των διαφόρων ε, επιτροπών μας. Η δική μας Επιτροπή Μηχανία μπορεί να υποστηρίξει η Επιτροπή μας τον όλο προβληματισμό σας και μάλιστα εν ώψη του, νέου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πράγματι, οι προπολογισμοί των κρατών μελών έχουν πληγεί ε, σε πολλούς τομείς και θα πρέπει από κοινού ε, να αντιμετωπιστεί το θέμα της άμυνας και όσον αφορά την ε, βιομηχανία των εξοπλισμών και τη σχετική επιστημονική έρευνα πρέπει να υπάρξει συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κράτη-μέλη που ε, προβληματίζονται και θέλουμε να κάνουμε συζήτηση, όχι να κάνουμε αξιολόγηση, αλλά ίσως και μαζί με τους βουλευτές των 100 μελών να δούμε τι συνέβη. Όσον αφορά τη συμφωνία που συνήθει μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, που ε, συνήψαν η συνθήκη για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων. Και κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει πολύ στην Επιτροπή Βιομηχανίας για τον βιομηχανικό τομέα και την τεχνολογική έρευνα και τα σχετικά προγράμματα. Αυτά τα δύο κράτη ενεντόπισαν 10 προτεραιότητες όσον αφορά την επικοινωνία μέσω δορυφόρων, τα drones, ε, τεχνολογία πολέμου, τα σκάφη, ηλεκτρονική τεχνολογία, προσωμιώσει, ε, διάφορα προγράμματα, έγκαιρος εντοπισμό ε, τρομοκρατικών δραστηριοτήτων κλπ. Υπάρχουν πολλέ δραστηριότητε που είναι δυτέ και στου δύο τομεί τον έφερε ε, και ο κύριος Γκάλερ, δηλαδή συνεργασία στρατιωτικού και πολιτικού τομέα. Άρα υπάρχει πεδίο συνεργασίας και χαίρομαι εκ των προτέρων που θα έχω δυνατότητα συνεργαστώ μαζί σας για να μπορέσουμε να υποβάλουμε τις καλύτερες δυνατές προτάσεις και να προτείνουμε πράγματα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Να προτείνουμε τα πιο χρήσιμα ε, για την όλη βιομηχανική βάση εξοπλισμού της Υπήρου μας. Ευχαριστώ, Σαν Πιέρ. Η κυρία Νικολάη, η αντιπρόεδρος μας, επιθυμεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ρουμανικά. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και χαίρομαι ιδιαίτερως ε, για τη συζήτηση αυτή. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον κύριο Γκάλερ και θεωρώ ότι θα καταλήξουμε σε πολύ ε, καλή επίσημη θέση. Μια στιγμή περιμένουμε να πατήσει το κουμπί γερμανική καμπίνα. Εντάξει. Το αποτέλεσμα μάλλον θα εξαρτηθεί από αυτά που έχουμε τώρα, από την τωρινή κατάσταση, αλλά και από τις επιθυμίες και τις προσδοκίες μας. Για να δημιουργήσουμε όμως μία βάση για την... Μία ε, βιομηχανική και τεχνολογική βάση άμυνα στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε πολιτική βούληση. Και βλέπουμε μέχρι στιγμής ότι ό,τι γίνεται, γίνεται σε εθνικό επίπεδο, όχι σε ευρωπαϊκό. Και από πολιτική άποψη υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του ευρωπαϊκού οράματος για κοινή πολιτική. Έχουμε κανόνες, διατάξεις, ε, θεσμικά όργανα, την συνθήκη της Λισαβόνας που αυξάνει τις αρμοδιότητές μας. Ζητάμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όλοι αυτοί οι κανόνες και οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται, δεν έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο ορατά και προφανή σε εθνικό επίπεδο και φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να προτιμούν εταιρικές σχέσεις και συνεργασία ε, και πολυμερή για την αμυντική βιομηχανία και έχουμε οργανισμούς και εταιρείε που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το μέλλον της ε, κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο στις Βρυξέλλες από το να θεσπίζουμε και να ιδρύουμε ε, θεσμούς και διατάξεις. Αν θέλουμε μια πραγματικά ενωσιακή πολιτική, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους υπάρχοντες μηχανισμούς. Εμένα με ενδιαφέρει ε, να αυξηθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Επίσης, ε, να έχουμε πιο συμβατούς κανόνες και προδιαγραφές για να καταλήξουμε σε κοινέ μονάδες παραγωγής. Γιατί μια και περικόπτονται συνέχεια οι προπολογισμοί και στον τομέα της άμυνας, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις επενδύσεις στον αμυντικό κλάδο. Ε, ακόμη και μιλούμε για διπλή χρήση, δηλαδή στρατιωτική και πολιτική, μη στρατιωτική και τις ε, διπλές αυτές τεχνολογίες. Επίσης θέλουμε κάποιους κανόνες ε, διαλειτουργικότητας και κάποιες κοινέ προδιαγραφές. Με κοινέ οικονομικές πολιτικές θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τα κράτη-μέλη από το να αγοράζουν συστηματικά εξοπλισμό μόνο από τρίτες χώρες. Γιατί θα πρέπει περισσότερο να αναπτύξουμε τη δική μας ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση στην άμυνα. γιατί μπορεί να έχουμε προγράμματα μακρόβια, αλλά νομίζω ότι ο βασικός μας πόρος ε, και ο βασικός μας, ε, η βασική μας προσπάθεια θέλουμε να βρούμε κάποια κοινά σημεία είναι και το σημαντικότερο φόρμα για τα θέματα αυτά είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Και έλπιζα η έκθεση να είναι λίγο πιο λεπτομεριακή και πιο ευρεία. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε επικοδομητικές προτάσεις ώστε να καταλήξουμε σε ένα όραμα που να είναι πιο συγκεκριμένο και από το και όχι μόνο θεωρητικό. Ευχαριστώ. Κύριο Ζέμκε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας. Βέβαια είναι η πρώτη συζήτηση που έχουμε με τα την παρουσίαση αυτή και δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα σχόλια που ήδη ακούσαμε. Θα ήθελα όμως ε, να επιστήσω την προσοχή σας ε, σε κάποια άλλα σημεία που δεν αναφέρονται, που κατά τη γνώμη μου όμως είναι σημαντικά. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από το πρώτο θέμα. Όταν μιλούμε για την βιομηχανία και την τεχνολογία, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη γνώμη μου, ε, είναι σημαντικό ότι στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, που δυστυχώς θα είναι ε, χαμηλότερο και πιο στενό από το προηγούμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ελιγμούς και κάποιες επιλογές. Θα πρέπει να αυξήσουμε τους πόρους για τις σύγχρονες τεχνολογίες και την καινοτομία αν δεν κάνω λάθος είναι 2 δισεκατομμύρια, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Πάντως στον τωρινό μας ε, προϋπολογισμό και στις τωρινές μας δημοσιονομικές προ... προοπτικές έχουμε γύρω στα 80 δις. Ενώ στον επόμενο προϋπολογισμό θα είναι 140 ε, δις. Έχουμε πολύ σημαντική περικοπή λοιπόν Βέβαια μπορεί να είναι δίκαιη αυτή η περικοπή λόγω της κρίσης, αλλά μας ε, οδηγεί αναπόφευκτα στην εξής ερώτηση, στον εξής προβληματισμό. Τα κοινοτικά μέσα, οι κοινοτικοί πόροι θα στηρίξουν ε, μόνο μελέτες ε, που καταλήγουν σε προϊόντα πολιτικού χαρακτήρα ή θα επιτρέψουμε την πιθανότητα από τα 40 και δισεκατομμύρια ένα τμήμα να αφιερωθεί σε στρατιωτικές τεχνολογίες. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι πολύ εύκολα στρατιωτικής χρήσης τεχνολογίες ε, ε, μπορούν να μετατραπούν σε πολιτικής χρήσης τεχνολογίες. Οπότε τα μέσα για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, κατά τη γνώμη μου, τα κοινοτικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για θέματα ασφάλειας και άμυνας, γιατί κάτι, κάτι τέτοιο θα δώσει μια νέα ποιότητα. Αλλιώς ε, ε, θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα χρηματοδοτήσουμε μόνο μελέτες ή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Νομίζω ότι ε, είναι σημαντικό επίσης να συγκεντρώσουμε τους πόρους και να κάνουμε κάποιες κοινέ ε, έρευνες. Τώρα έχουμε κάποια βασικά προβλήματα σήμερα. Όχι μόνο ότι μειώνονται οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς με τον κύριο Ζαλεύσκη ανήκουμε ε, καταγόμαστε από μια χώρα που δεν κάνει περικοπές στις αμυντικές δαπάνες, γύρω στο 2% του ΑΕΠ, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες που δυστυχώς περικόπτουν τις αμυντικές δαπάνες και μάλιστα μειώνονται και τα κονδύλια προς τις νέες τεχνολογίες. Φαίνεται ότι κάνουν άλλες επιλογές τα κράτη-μέλη. Οπότε αυξάνεται όλο και μεγαλύτερα, το, αυξάνεται και περισσότερο το χάσμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και με άλλες αναδυόμενες χώρες όπως η Κίνα ή άλλες που αφιερώνουν πολύ περισσότερα στις αμυντικές τους δαπάνες. Πιστεύω ότι η άμυνα θα πρέπει να αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα. Αυτή είναι η δεύτερη μου παρατήρηση. Τώρα, τρίτη παρατήρηση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε στο υλικό αυτό να κάνουμε έναν απολογισμό κάποιων περιττών δαπανών που κάνουμε στην ε, Ευρώπη, γιατί έχουμε ε, διάφορα προγράμματα για τα τεθωρακισμένα ή για μελέτες για τα υποβρύχια. Ε, τεράστιες δαπάνες γίνονται για αυτά τα προγράμματα, αλλά φαίνεται ότι στην Ευρώπη η παραγωγή είναι πολύ πιο ακριβή από ό,τι αλλού. Θα πρέπει λοιπόν και αυτά τα θέματα ίσως να τα επισημάνουμε στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Merci, Madame Kronberg. Ευχαριστώ, κυρία Κρόμπεργκ. <clears throat> Is... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Το πρόβλημα ήταν από όταν δημιουργήθηκε το πριν από 15 χρόνια ε, δεν συνέβησαν πολλά. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή τεχνολογική βιομηχανική βάση για την άμυνα. Ή αυτή η βιομηχανία βασίζεται στην γαλλική βιομηχανία, βρετανική βιομηχανία, φιλανδική ε, βιομηχανία, το τοπίο το αμυντικό στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικότητα, ε, υπερβολική παραγωγή ε, και πολύ εθνικιστική προσέγγιση. Η συνεργασία δεν είναι καθόλου καλή και η δυνατότητα του ΝΑΤΟ και της ΚΕΠΑ έχει πάρα πολλά κενά. δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι μπαίνουμε σε ανταγωνισμό με τη ΣΥΠΑ. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να δούμε ποιε είναι οι συγκεκριμένε δυνατότητε που υπάρχουν. Ποιε είναι οι γνώσει που υπάρχουν. Και ποια τα πλαίσια για ευρωπαϊκή συνεργασία. Όχι σε εθνικό επίπεδο συνεργασία μεταξύ κρατών. Και δεν θέλουμε να αναπτύσσονται οι τεχνολογίε σε εθνικό επίπεδο. Για του πρασίνου ε, πρέπει να γίνουν ε, μεγάλε διαθωτικέ αλλαγέ Και ε, όπως έχει η κατάσταση τώρα, είναι πολύ δύσκολο να επενδυθούν νέοι πόροι σε αυτό το τομέα. Η κυρία Λούζιν έχει το λόγο. Ο κύριος Γκάλα ε, στην εισαγωγή του αναφέρθηκε κυρίως ε, ε, στους στόχους και η κυρία Νικολάη αναφέρθηκε και αυτή σε αυτό. Και εγώ την πρώτη μου ερώτηση θέλω να την κατευθύνω προς αυτό το θέμα. Δηλαδή, τελικά, αν υπάρξουν διαδικασίες αναδιάρθρωσης, αν υπάρξει ισχυρότερη τεχνολογία και ε, βιομηχανική βάση, τότε ποιος θα καθοδηγήσει αυτή την εξέλιξη. Η κυρία Νικολάη μίλησε για την ενίσχυση του Οργανισμού Άμυνας, δηλαδή αυτή η διαδικασία θα πρέπει να καθοδηγηθεί από αυτόν τον οργανισμό ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αν καθοδηγηθεί η εξέλιξη αυτή από την Κομισιόν, ερωτώ εγώ, ποιες είναι οι απόψεις του εισηγητή για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτής της διαδικασίας. Κατόπιν ε, διάφοροι ομιλητές ε, αναφέρθηκαν ε, στο θέμα της χρηματοδότησης, δηλαδή στο ερώτημα με ποιο τρόπο ή σε ποιες ποσότητες εκταμιεύονται κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση αυτής της διαδικασίας ή ποια είναι τα κονδύλια που επενδύονται στην έρευνα εγώ λοιπόν, ε, όπως ε, ερμηνεύω ε, το άρθρο 41 παράγραφος 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση αυτής της εξέλιξης δεν μπορεί να γίνει με κοινοτικά κονδύλια. Και θα ήθελα να ακούσω την άποψη του εισηγητή για αυτό το τόσο περίπλοκο θέμα, όπως επίσης και την άποψη των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ θα κλείσουμε αυτό το γύρο ανταλλαγής απόψεων που είναι προκαταρκτικό στάδιο. Ε, Μίκαελ, δεν ξέρω αν έχεις αποσθέσει κάτι. Σα ε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, τοποθέτηση. Χαίρομαι πολύ για τη συνεργασία με την Επιτροπή Βιομηχανίας, με όλους τους συναδέλφους. Τα θέματα που ετέθησαν ήταν πολύ σημαντικά. Ας πούμε το θέμα της διαλειτουργικότητας. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο καθιστά σαφές ότι αναζητούμε ε, τρόπους ενοποίησης ε, των αμυντικών προμηθειών και εκτός Ευρώπης. Ο στόχος ε, πρέπει να είναι να αποφύγουμε τη διασπάθηση κονδυλίων. Ο στόχος πρέπει να είναι μέσα από κοινού ε, διαγωνισμούς να εξοικονομούμε κονδύλια, να διασφαλίζουμε τη διαλειτουργικότητα και επίσης στο μέλλον να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια που είναι όλο και λιγότερα ε, για τέτοιου είδους ε, αγορές εξοπλισμών. Το καθοριστικό ερώτημα που ετέθη είναι ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν για τη συνεργασία. Για μας το καθοριστικό ερώτημα είναι κατά πόσον είμαστε σε θέση ε, την ασφάλεια των ε, προμηθειών ε, να τη χρησιμοποιήσουμε για την εφαρμογή της πολιτικής μας. Δηλαδή σημαντικό είναι τι θέλουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες είναι οι αποφάσεις μας και όσον αφορά τις αποφάσεις μας έχουμε τη βάση να είμαστε αυτόνομοι. Γιατί αν εξαρτώμεθα απ' έξω, μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω αν θα μπορούμε ε, να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια. Αυτό για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το να ξέρουμε δηλαδή ότι για στρατιωτικές ε, και πολιτικές επιχειρήσεις, να είμαστε σε θέση να ε, ολοκληρώσουμε τις επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, ποιος θα καθοδηγήσει τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης. Κοιτάξτε, ας είμαστε ρεαλιστές. Εδώ μιλάμε για κατανομή αρμοδιοτήτων. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, δηλαδή για θέματα κοινή αγοράς. Νομίζω όμως ότι η διαδικασία της ε, αναδιάρθρωσης ε, μάλλον θα λάβει χώρα περισσότερο υπό την καθοδήγηση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Χωρίς αυτήν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρόκειται για συντονιστικές αρμοδιότητες ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Και όσον αφορά τη νομική βάση, ε, στον ερευνητικό τομέα μπορούμε να χρησιμοποιούμε προϊόντα διπλής χρήσης, dual use. Εγώ τη νομική βάση έτσι τουλάχιστον την ερμηνεύω. Βεβαίως ε, μπορούμε να εφαρμόσουμε και άλλη πολιτική με βάση τις συνθήκες, ότι εξυπηρετεί το στόχο, θα πρέπει να μπορούμε να το υλοποιούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ζαν Πιεροντή, θέλω να πω εν συντομία ότι λησμόν σας πω ότι επεξεργαζόμαστε το θέμα του διαστήματος με το πρόγραμμα Γαλιλαίος που είναι σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ούτω ώστε το σήμα να είναι εξάρτητο από το αμερικανικό σήμα και με εφαρμογέ στατιστικέ προφανώ οι οποίε προβλέπονται στο όλο διατακτικό, καθώ και με το Κοπέρνικο, στο παλιό πρόγραμμα GMS. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι άκουσα προσεκτικά τι διάφορε παρεμβάσει των διαφόρων βουλευτών και των πολιτικών ομάδων που καταδεικνύει τη χρησιμότητα που έχει να συνταχθεί αυτή η έκθεση και χαίρομαι και το λέω ξανά που θα συνεργαστώ με τον συνάδελφο Γκάλερ υπό ε, συνθήκες που θα καθορίσουμε ε, μαζί από κοινού στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 50. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Λοιπόν, θα πρέπει να είστε μελετηροί, διότι θα γίνει μια εξέταση του πρώτου κειμένου στις 18 Σεπτεμβρίου και το θέμα, επαναλαμβάνω, ότι είναι στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου και θα είναι πολύ καλό το Κοινοβούλιο πάνω σε αυτό να μπορεί να έχει μία θέση όσο πιο ενωμένη γίνεται το φθινόπωρο πριν από τη συνεδριάση τη σύνοδο αυτή του τέλους του έτους, ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας. Ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση και πάμε στο επόμενο σημείο. Καλή ψηφοφορία, καλή δουλειά. Με καλή επόμενο σημείο είναι πιο πρωτότυπο όσον αφορά τη σύνθεση και την ουσία, αλλά εξίσου ενδιαφέρον και από, πλευρές, από πολλές πλευρές ε, άπτεται των θεμάτων που συζητήσαμε. Ήθελα λοιπόν να έχουμε ανάμεσά μας επιφανείς εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, οι οποίοι ε, επεξεργάστηκαν συστάσεις για μια λευκή βίβλο για την ασφάλεια και άμενα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Νομίζουμε ότι αυτό το έργο, αυτή η δουλειά ε, είναι πολύ σημαντική και θεώρησα ότι θα χρειαζόταν να ρίξουμε τους προβολείς επιτροπής μας σε αυτό το έργο διότι αυτή η Επιτροπή πρώτα απ' όλα από καιρού μέσω των διαφόρων ετησίων εκθέσεων ζητά την επεξεργασία λευκής βίβλου για την ασφάλεια και την άμυνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαιρετίζω και την παρουσία του Κάλφον Βογκάου, τον προκάτοχό μου χαιρετίζω, που όταν ε, μου, έδωσε τη σκητάλη είχε αναφέσει αυτό το στοιχείο. Εγώ δεν είμαι ένθεμος υποστηριχτής αυτού του στοιχείου διότι το όλο εγχείρημα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες ε, μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων όσον αφορά τι διάφορε προτεραιότητε που πρέπει να επιτευχθεί η συμφωνία και ομολογώ ότι ήμουν κάπω διστακτικό μετά κατά τη διάρκεια τη θητεία των καθηκόντων μου. Διαπίστωσα ότι είχε απόλυτο δίκιο και ότι αν το Κοινοβούλιο δεν επέμενε ούτω ώστε να υπάρξει μια μεθοδολογία όσον αφορά τη στρατηγική προσέγγιση, κανεί άλλο θεσμικό δεν θα το έκανε στη θέση του. Σε αυτή την περίπτωση το κάνουμε υπενθυμίζουμε μεγάλη υποστήριξη το θέμα κάθε χρόνο και είμαι πολύ ευτυχής που επιφανής πανεπιστημιακή με ένα παρελθόν όμως ε, πρακτικής εμπειρίας, πολύ αξιοσημείωτο, ε, έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό, κυρίως φέτος, διότι είναι το περίφημο συμβούλιο θα λάβει χώρα στο τέλος του έτους. Λοιπόν, να συνεννοηθούμε, δεν διεκδικούμε και δεν περιμένουμε αρχική κρατών και κυβερνήσεων που θα συνεδριάσουν το Δεκέμβριο για να μιλήσουν για την πολιτική της άμυνας, να υιοθετήσουν εκείνη την ημέρα μια λευκή βίβλο. Περιμένουμε όμως τουλάχιστον κάποια μηνύματα, κάποια σημάδια, ελάχιστα αν θέλετε, κάποια μηνύματα που θα δείχνουν ότι αυτή η μεθοδολογία επιτέλους θα ριζώσει στις όλες τις διαδικασίες που θα ξεκινήσουν μετά τον ε, Δεκέμβριο. Ε, πρέπει να πω ότι προκαταρτικές συζητήσεις που είχατε εσείς και εμείς με τα διάφορα θεσμικά όργανα, εθνικά ευρωπαϊκά, βλέπουμε τις δυσκολίες που δημιουργεί η συζήτηση. Δηλαδή όλος ο κόσμος έχει επίγνωση ότι χωρίς στρατηγικό όραμα, ανανεωμένο διότι στρατηγικό όραμα υπήρχε, δεν λησμονώ τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν χρησιμίστες το 2003 και αναθεωρήθηκαν το 2008, αλλά βλέπουμε την ανάγκη υπάρχει για ανανέωση του στρατηγικού προβληματισμού, να ανοίξουν προοπτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο στρατηγικό περιβάλλον, και βλέπουμε ότι ακόμα και είναι μεγάλος ο πειρασμός και αν οι ανάγκες γίνονται αισθητέ, και πολλοί αισθητέ, υπάρχει δισταγμό, σοβαρό δισταγμό σε πολιτικό επίπεδο για να ξεκινήσει η συζήτηση. Υπάρχουν φόβοι, θα έλεγα, φόβοι μήπω ξεφύγει η συζήτηση προ ανατολικά, προ νότο για νέε απειλή και θα έχουμε πρόβλημα να ιεραρχήσουμε τι προτεραιότητε. Περί αυτού πρόκειται. Και για αυτού όπω εγώ που ζητούμε το άνοιγμα τη συζήτηση για τη μεθοδολογία τη Ευχή Βίβλου, ξεπερνά την απλή αποτίμηση των απειλών, απλή εκτίμηση των νέων διεθνών φορέων, μη απογραφή των συμφερόντων των ευρωπαϊκών ή του δυναμικού που διαθέτουμε, πραγματικά πρόκειται για κάτι άλλο, για ένα νέο στατηγικό προβληματισμό πρόκειται που επιβάλλεται και χαίρομαι πολύ που υποδέχομαι εδώ για την παρουσίαση των συστάσεων και των εργασιών. Πολλούς ε, διακεκριμένους του κυκλημένους, κάποιος θα έρθει αργότερα δυστυχώς. Εγώ θα έχω φύγει τότε δυστυχώ. Η συζήτηση όμω θα μπορούσε παρόλα αυτά να συνεχιστεί. Λοιπόν, θα ακολουθήσουμε τη σειρά, διότι ξέρω ότι οι εργασίε είναι πολύ καταστασμένε. Έχουμε τον καθηγητή Σεμινατόρε, γνωστό εδώ, ο οποίο προεδρεύει το Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και είναι στη βάση, βρίσκεται στη βάση τη όλη πρωτοβουλία. Και πολύ ε, πρώιμα, πολύ αρχικά ανέλαβε αυτό το καθήκον. Τον ευχαριστώ που μα ενημέρωνε για τι εξελίξει των εργασιών και θα μιλήσει πρώτος. Έχουμε τον στρατηγό Έρικ Τελαρία που θα επιμένει πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε κάποιες δυνατότητες, κάποια προγράμματα και συγκεκριμένες προσπάθειες που θα πρέπει να καταληθούν σε ευρωπαϊκή επίπεδο. Έχουμε και τον πρέσβη Μορέλ που τον έχουμε υποδεχτεί πολύ συχνά σε αυτή την επιτροπή μας υπό άλλη ιδιότητα για τις εργασίες του που έκανε του ειδικού εκπροσώπου στην Κεντρική Ασία για την κρίση στην Γεωργία και, και ο Μπίτερλιχ, ο πρέσβης ο κ. Μπίτερλιχ έχει έρθει που ήταν διπλωματικός σύμβουλος του καγκελαρίου Κολ και που θα ολοκληρώσει την όλη παρουσίαση. Αυτά εν συντομή, αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου θα διεξαχθεί αυτή η συζήτηση, είναι αρκετά πρωτότυπη, αλλά θέλω να επενθυμίσω, έχει πραγματικά τη θέση της στις όλες προπτικές ε, που δημιουργούνται εν ώψη του Συμβουλίου του τέλους του έτους και χρειάζεται μια δημόσια συζήτηση ε, για το πρόγραμμα αυτό και για τη συζήτηση που λάβουν χώρα. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Λοιπόν, καθηγητά, κύριε Σεμινατόρα, είχετε το λόγο. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι Ευρωβουλευτέ, η Μονάδα Στρατηγικής Σκέψης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων σας υποβάλλει τις ε, συστάσεις της για μια λευκή βίβλο για την άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέσσερις ανεξάρτητες προσωπικότητες από τις 16 που συνέβαλαν στην κατάρτιση αυτών των συστάσεων θα σας εξηγήσω το σκοπό, τη θεματική διάρθρωση, τις ε, θεσμικές και στρατηγικές συνέπειες ε, και κάποιες γενικές επιπτώσεις. Καταρχήν γιατί προτείνουμε μια λευκή βίβλο γιατί βρίσκεται στην, θέτει στο επίκεντρο ε, του ενδιαφέροντος, ε, της προσδοκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια αυξημένη ανάληψη ευθύνης ε, στην Ήπειρο, στις γειτονικέ χώρες αλλά και στον κόσμο. Επίσης, προτείνει τον καθορισμό διπλωματικών και στρατιωτικών στόχων που στα πλαίσια της κοινή ε, επιτροπή ε, Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, που νομίζω στα πλαίσια της διεθνής μας θέση είναι πολύ σημαντικό. Είναι υπέρ μια διπολικής προσέγγισης, θέλει να κρατήσει την αυτονομία της Υπήρου ε, και είναι κατά μια, ενός αφοπλισμού της Ευρώπης έναντι σε μια αυξανόμενο, αυξανόμενο εξοπλισμό της Ασίας. Το έγγραφο που προτείνουμε θεωρεί ότι το εσωτερικό πολιτικό πλαίσιο και η διεθνή συγκυρία αλλά και το περιβάλλον ασφάλειας είναι σημαντικά διακυβεύματα και προκλήσεις ε, στα οποία θα πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που χαρακτηρίζεται από 27 διαφορετικά συστήματα λήψη αποφάσεων και χαρακτηρίζονται μερικές φορές από διάσταση απόψεων. Θεωρεί ότι θα πρέπει να ε, υιοθετηθεί μια κοινή προσέγγιση απέναντι στις κρίσεις ε, ε, και τις απειλές ε, που δημιουργούνται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθεί η συνεργασία σε βιομηχανικό επίπεδο, να ενισχυθούν οι ικανότητες σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και προτείνει μια στρατηγική κοινή, διαφοροποιημένη και σφαιρική. Μια στρατηγική με όλη το νόημα του όρου. Και το κείμενο που σας προτείνουμε είναι ένα ακαδημαϊκό έγγραφο που προσπαθεί να συνδυάσει εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια συμφέροντα. Στόχο έχει να προσδιορίσει τους, τις φιλοδοξίες, τους πόρους και την πολιτική βούληση της Ένωσης, ε, κάνοντας μνήα της κοινοτική συνοχής και της υπάρχουσας θεσμικής ε, διάρθρωσης. Επίσης, ε, κρούει το κόδωνα το κινδύνου σε ό,τι αφορά το χάσμα στον, στον κυβερνοχώρο και στα τεχνολογικά θέματα μεταξύ Ευρώπης ε, και Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης και Κίνας. Τώρα, για ποιους λόγους συντάξαμε τη Λευκή Βίβλο θεωρούμε ότι αν στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποκτήσει μια πολυπολική στρατηγική και μια ε, διπλωματική παρουσία στις διάφορες ζώνες του κόσμου και αν η στρατηγική της αυτή δεν είναι αρκετά διαφοροποιημένη από θεσμικό και γεωπολιτικό επίπεδο, η Ευρώπη θα περιθωριοποιηθεί στον 21ο αιώνα. Αν η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προωθήσει μία επανάσταση στα πολιτικά και στρατιωτικά τεκτενόμενα θα εξαφανιστεί από τους βασικούς εταίρους. Γι' αυτό η, στρατηγική, η πολυπολική στρατηγική είναι επιτακτική ανάγκη. Τώρα έχουμε το συμπέρασμα αυτό που στηρίζεται σε βασικά κριτήρια. Καταρχήν θα πρέπει να αντιληφθούμε το σχετισμό δυνάμεων παγκοσμίω και η θα πρέπει να δούμε, ε, ε, να λάβουμε υπόψη τους τρεις στόχους, ε, τον, τον διπλωματικό, τον βιομηχανικό και τον αισθητικό. Θα πρέπει να αποφύγουμε, να αποφύγουμε τη βαλκανοποίηση και επίσης να λάβουμε υπόψη το σχετισμό δυνάμεων μεταξύ των διαφόρων εταίρων. Γιατί υπάρχουν κάποιες επικίνδυνες ζώνες που ήταν ανέκαθεν επικίνδυνες γιατί δημιουργούν μια αναποφασιστικότητα και στρατηγικό κενό που με μερικές φορές οδηγούν σε απρόβλεπτα αποτελέσματα. Άλλη συνθήκη είναι η επανισορρόπηση της σχέσης μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών εταίρων εντός του ΝΑΤΟ και δεδομένη τη ε, στρατητική και πολιτική συνεργασία, και θα πρέπει να δούμε την περιφερειακή ε, συμμαχική ε, στην Ευρώπη πολιτική και την έννοια της παγκόσμιας ασφάλειας. Επίσης, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο σε θέματα εξοπλισμού προκειμένου να ενισχυθεί η βιομηχανική δομή στα πλαίσια μιας αγοράς άμυνας που θα είναι ειδική και δεν θα θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα εθνικά μοντέλα άμυνα στι ευρωπαϊκέ φιλοδοξίε και εξασφαλίζοντα προνομιακή πρόσβαση τη ευρωπαϊκή βιομηχανία στα ετήσια προγράμματα καθώ και τα προγράμματα έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Και τέλο, πρόθεση τη Ευρώπη ω παγκόσμιο φορέα και παγκόσμια δύναμη. Κάτι που προποθέτει μια, μια ενοιολογική επανάσταση και μια εξέλιξη στα πολιτικά και στρατηγικά θέματα λήψη υπόψη την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα λέιζερ, δορυφορική παρακολούθηση. Αυτά είναι βασικά σημεία που χαρακτηρίζουν ε, τους παγκόσμιους ε, φορείς, τις παγκόσμιες δυνάμεις. Επίσης, η πολυπολική προσέγγιση του παγκόσμιου συστήματος καταλήγει ε, κατά ανάγκη και λογικά και κατά συνέπεια στον προσδιορισμό μια πλανητική στρατηγική που θα, έχει, θα στηρίζεται σε ένα τριγωνικό χαρακτήρα. Η στρατηγική αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο ε, τη ε, στρατηγική ασφάλεια ε, που προτείνει η Λευκή Βίβλο και ε, λαμβάνει τρει μορφέ και έχει χαρακτήρες hard, smart και soft. Ας κυρίσω από το σκληρό χαρακτήρα. Στρατηγική hard ε, σφαιρική ε, και ασχολείται με τα ζωτικά συμφέροντα. Παρακολουθεί τη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την διπολικότητα στην πολυπολικότητα και προσδιορίζει μακροπρόθεσμους στόχους για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στόχο η χάρτη στρατηγική έχει την εξασφάλιση της σταθερότητας του διεθνού συστήματος καθώς και την ε, προστασία της Ένωσης από πολύμορφες απειλές, εσωτερικές ή εξωτερικές διεθνείς, που ε, θέτουν σε κίνδυνο την ισχυρή της θέση και την επιβίωσή της. Ε, η smart στρατηγική, η έξυπνη στρατηγική, ε, λαμβάνει υπόψη τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πολυπολική διάρθρωση και θα πρέπει φυσικά να προσανατολίζεται από την γάλλο-γερμανική ηγετική θέση που θα προσαρμόζεται όμως στα ευρωπαϊκά δεδομένα η πολιτική και στρατηγική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναχθεί σε πλανητική κλίμακα, σε αυτή του σχετισμού δυνάμεων του 21ου αιώνα. Επίσης θα πρέπει να έχει και προληπτικό χαρακτήρα. Ε, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την ε, πολυπολική στρατηγική ως στρατηγική επανισορρόπησης και παγκόσμιας προσαρμογής ε, με ενεργό proactive χαρακτήρα. Επίσης, ε, να βάλουμε υπόψη τις μόνιμες ε, συμμαχίες, ε, την χρήση της βίας και την αρχή της, αυτο... της στρατηγικής αυτονομίας. Είναι προληπτική στρατηγική σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τώρα, από στρατηγική άποψη, καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δράσεων, συμβατικών, βαλιστικών, τεχνολογικών, πυρηνικών, δορυφορικών, της ασφάλειας του κυβερνοχώρο και βιομηχανικών. Και επίσης συγκεντρώνει και τις ε, λειτουργίες συντονισμού. Τώρα η στρατηγική SMART, ευφυή e, στρατηγική όπως λέει ο, το ΝΑΤΟ και τη λέμε SMART γιατί βρίσκεται μεταξύ της hard και της soft στρατηγικής, της ε, ε, σκληρής και της ήπιας. Η ευφυή e στρατηγική είναι μεικτή, διακρατική και αφορά την συλλογική ασφάλεια, τις περιφερειακές συγκρούσεις και τις μεγάλες κρίσεις γειτονίας ή του δεύτερου κύκλου που διακυβεύουν τα γειτονικά συμφέροντα της Ένωσης στα πλαίσια των ε, ε, κοντινών δράσεων. Πρόκειται για μια σταθεροποιητική δράση. Η πρώτη δράση είναι της επανισορρόπησης, η δεύτερη δράση, η στρατηγική SMART, είναι της ε, σταθεροποίησης. Θα πρέπει να λάβει υπόψη διάφορα στοιχεία, κοινωνικο-οικονομικά, κατασταλτικά, προληπτικά, δημοσιονομικά, ενεργειακή πολιτική και κοινωνική πολιτική και τα συνδυάζει στα πλαίσια δογματικών κατηγοριών που θα πρέπει να είναι γενικές και ως τέτοιες συγκεχημένες δημιουργούν πηγή δράσης και λαμβάνει τη μορφή μιας στρατηγικής διαχείρισης της κρίσης μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας, μιας ιεράρχησης των εθνικών συμφερόντων, της διασφάλισης των συνόρων της Ένωσης, της κοινή χρήση των πόρων αλλά κυρίως και των ευθυνών η soft στρατηγική, η ήπια στρατηγική, η πολιτισμική στρατηγική είναι η βασική στρατηγική της ε, ε, Ευρώπης που λαμβάνει ένα συμβολικό χαρακτήρα και εκεί είναι που κερδίζονται ή χάνονται οι μάχες της ιστορίας. Ο συμβολικός της χαρακτήρας της εξασφαλίζει μία αναφυσβήτητη και κοινή νομιμοποίηση. Είναι φιλοπολιτιστική και ε, συνάδει με την εμπορική και την νομική στρατηγική και κυρίως πρόκειται για μια στρατηγική που, δίνει, ε, που έχει υπαρξιακό χαρακτήρα, χαρακτήρα ταυτότητας και στηρίζεται σε, ένα, σε μια πρόκληση και εκεί το μεγαλείο μιας ιδέας απέναντι στο έθνος είναι θέματα ε, νοητικής προσπάθειας αλλά και κοινή ανάληψης ευθυνών. Η στρατηγική αυτή αφορά μια κοινότητα ε, πεπρωμένου και χαρακτηρίζεται από τις θεμελιώδεις αξίες και τα μεγάλα τις οράματα για τον κόσμο. Οπότε η προσέγγισή μας δίνει μια πρώτη απάντηση στην ανάλυση της παρούσας κατάστασης, αλλά και της, του γενικού πλαισίου και προτείνει πολύ σημαντικές συστάσεις. Και οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας χρήζουν ενιαίες απαντήσεις που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, και καθιστούν τη στρατηγική και πολιτική ενότητα της Υπήρου πιο σημαντική από ποτέ. Για να προωθηθεί η ειρήνη και να, και να προετοιμάσει το μέλλον θα πρέπει να δημιουργήσουμε ασφάλεια και να χτίσουμε την ασφάλεια και για μας αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ καθηγήτα. Ζεράρ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για να δώσω συνέχεια στις πρώτες πτυχές όσον αφορά το θεωρητικό στοιχείο, πήραμε και την πρακτική πλευρά, λαμβάναμε υπόψη την επιχειρησιακή ε, πτυχή της ε, επαναπρόθεσης της ΚΕΠΑ εν ώψη των μονίμων διεθνών κρίσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έναντι των οποίων η πολιτική βούληση να μπορεί να υπάρξει στήριξη σε αποτελεσματικά εργαλεία και οικονομικά βιώσιμα αντιμετωπίζονται δύο ευαίσθητοι τομείς που είναι ε, οι πληροφορίε για τον κυβερνοχώρο και διάφορε άλλε πτυχέ που ίσω να ενδιαφέρουν τι προπαρασκευαστικέ κρατήσει του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πληροφορίε. Η επιτυχία τη εξωτερική πολιτική αφορά τη συλλογή και εκμετάλλευση αξιοπίστων πληροφοριών. Πρόσφατα είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση παρενέβη σε κάποιε περιοχέ και χρειάστηκαν ε, χρειάζεται καλό εξοπλισμό συλλογή πληροφοριών, καταρτισμένο προσωπικό, χρειάζεται διαλειτουργικότητα απαραίτητα και χρειάζεται συνεχής επαλήθευση των πηγών των πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές είναι κάτι που συνήθως είναι στα χέρια των ε, κρατών και χρειάζεται σχεδιασμό για τη συλλογή των πληροφοριών και αυτό είναι πολύ απαραίτητο για το μέλλον. Χρειάζεται μεγάλη πειθαρχία, πρέπει να γίνονται συγκεκριμένε προσπάθειες γι' αυτό. Και όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, και την έρευνα και τεχνολογία, τη βιομηχανική παραγωγή και την κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού. Τρει στοιχέ, κατά την άποψή μα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προτεραιότητα λόγω του κρίσιμου χαρακτήρα που έχουν. Πρώτον, οι πρόσφατε πληροφορίε που είδαμε, τα μαθήματα από τα Βαλκάνια, το Αφγανιστάν στην Αφρική, ε, επί εδάφου, αέρος και θαλάσσης, δείχνουν ότι χρειάζεται να έχει κανεί αξιόπιστες πληροφορίε σε πραγματικό χρόνο για σχεδιασμό και διεξαγωγή αποστολών και θα πρέπει ε, αυτές οι αποστολέ πραγματοποιούνται με μια επανδρομένα οχήματα, drones. Κάποια κράτη-μέλη ε, πρέπει να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν κατεπηγόντω κάποια μέσα αντιμετώπιση ανάγκη τη Ένωση. Για και καμιά φορά λείπει εξοπλισμό και μόνο τρίτε χώρε μπορεί να δώσουν το εξοπλισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει παραλύσει η Ευρώπη στον τομέα. Υπάρχει δυνατότητα τεχνολογική, υπάρχουν γνώσει εντό των επιχειρήσεων για, τα, για τον απαραίτητο εξοπλισμό. Παράλληλα, σε ένα πλαίσιο όπου εξωτερική ασφάλεια και εσωτερική ε, αλληλεκαλύπτονται, η δυνατότητα των μη επανδρομένων οχημάτων καλύπτει ανάγκε. Ε, Κυρίω να στραφούμε κατά τη μεγάλη εγκληματικότητα, που οδηγεί σε ε, ένοπλα κινήματα και αντιμετωπίζονται στο, στα, στα πεδία της μάχης. Λοιπόν, θα πρέπει στο Συμβούλιο να, να προωθηθεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα drones μη παδρομένων χημάτων που να μπορούν να έχουν μακρά διάρκεια πτήση σε ψηλό επίπεδο και να χρησιμοποιούνται διτά. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό στόλο αυτών των μη επανδρομένων οχημάτων. Δεύτερον, αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών που διαδέχθηκε το ε, αυτό εδράζεται επί της ροής πληροφοριών που δέχεται να δώσει, δέχονται να δώσει τα κράτη-μέλη. Ο συντονιστή πληροφοριών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, στην προσπάθεια καταβολή τρομοκρατία μπορεί ε, να είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Σε μεταγενέστερη φάση θα πρέπει να έχουμε υπηρεσία Ευρωπαϊκή Πληροφοριών που θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασία των στοιχείων και συντονισμού στον τομέα που αφορούν εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια τη Ένωση. Τρίτο σημείο. Όσον αφορά την κατάρτιση και την παιδεία, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα τελειοποίηση όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών για του ειδικού του τομέα μπορεί να δημιουργηθεί, παραδείγματο χάρη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κολεγίου για την ασφάλεια τη και την άμυνα, συμπληρώνοντα την εθνική κατάρτιση, βέβαια, αυτό ξυπακούεται. Σχετικά με αυτό, δεν θα πρέπει να μελούμε τα συνέπειε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, υπό τον όρο ότι οι δυσκολίε πολιτικέ που επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ κάποιων μελών των δύο οργανισμών να μπορούν βέβαια να ξεπεραστούν. Δεύτερη πτυχή που θα θέλαμε να εξετάσουμε είναι της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας. Στον ευαίσθητο τομέα αυτό που είναι η κυβερνοασφάλεια και η κυβερνοάμυνα και που ήδη τον Νοέμβριο του 2012 συζητήθηκαν τα θέματα, ε, άλλαξε η κατάσταση μετά την εμφάνιση του εγγράφου για τη στρατηγική της Ένωσης στον τομέα. Λοιπόν, ο κυβερνοχώρο οδηγεί σε πρόοδο, αλλά δημιουργείται και νέοι κίνδυνοι για αυτόν, κυρίω για τι κρίσιμε εθνικέ και κοινοτικέ υποδομέ. Αλληλένδετο με το θέμα των πληροφοριών που προαναφέραμε, ο κυβερνοχώρο είναι ένα θέατρο επιχειρήσεων εικονικό όπου ο αντίπαλος δεν έχει πρόσωπο και μπορεί να διεισδύσει με πιο περίπλοκους τρόπους σε ένα πλαίσιο νομικό όπου η ειρήνη, κρίση, πόλεμος ε, διαχωρίζονται με πολύ ακαθόριστες διαχωριστικές γραμμές. Η Ένωση άρα δεν έχει άλλη εναλλακτική μου φαίνεται παρά να επιμείνει επί μιας ευρωπαϊκής κυβερνοστατηγικής ή κυβερνοαμήνης και καταπολέμης εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο και θα πρέπει να γίνουν προσπάσει σε αυτού του τομείς. Και είναι αλληλένδετα αυτά. Θα πρέπει οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορεί να προστατευτούν μέσω καλύτερη ενημέρωση για του κίνδυνου που διατρέχουν και θα πρέπει εκεί να υπάρχει ένα συντονιστή για την κυβερνοασφάλεια που θα ασχολείται με τον εξοτολογισμό των δράσεων της έρευνας, της βιομηχανικής πολιτικής και της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής, που πολύ συχνά αυτά αντιμετωπίζονται κατακαιρμισμένα από τους θεσμικούς φορείς και τα Το πρόγραμμα λοιπόν προτείνει τέσσερις πυλώνες, συνοχή, που συμφιλιώνει την ελευθερία με την ασφάλεια και επιτρέπει την αρμόνιση των πολιτικών που βασίζονται στα νομικά εργαλεία που υπάρχουν και τα μελλοντικά εργαλεία. Δεύτερο, συντονισμό που είναι προπόθεση για την επιτυχία που θα βασίζεται στη διακυβερνητική προσέγγιση, θεσμική προσέγγιση, συνεργασία μεταξύ 100 μελών, συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψει που είναι δαπανηρέ ο συντονιστή για την κυβερνοασφάλεια θα μπορεί έτσι να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Η Πολιτική Επιτροπή και η Επιτροπή Ασφάλεια, οι επιτροπέ αυτέ μπορούν να καθορίσουν σε μια επαφή επιφορτισμένη την παρακολούθηση τη ασφάλεια και τη κυβερναμίνη. Τέλο, η συνεργασία που ταιριάζει με τη συνοχή και συντονισμό συνεπάγεται μια ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 100 μελών επιθελοντική βάση σε σχέση με άλλε σχετικέ δομέ όπω το Κέντρο Αριστεία του ΝΑΤΟ που αφορά την κυβερνοάμυνα, την Ευρωπόλ ή την ΕΝΙΣΑ. Τώρα, όσον αφορά το δυναμικό που υπάρχει, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα διάφορα επιστάμενα προγράμματα, υπό αυτά που τελούν υπό εξεργασία, δίνοντα τα οικονομικά και ανθρώπινα μέσα για να μπορέσουν να πετύχουν το στόχο. Θεωρητικά, όσον αφορά τι μελέτε που διεξάγονται στα στρατηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την τεχνολογική κατάρτιση, όσον αφορά τι πληροφορίε και την επικοινωνία και τα συστήματα ασφαλεία, όσον αφορά τη διάδοση των πληροφοριών, σε επιχειρησιακό επίπεδο μέσω τη αντιμετωπίση του ΣΕΡΤ, της, ομα, της, ε, της ομάδας κατεπίγους παρέμβασης στην πληροφορική και θα πρέπει να υπάρχει πτυχή άμυνα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης Κυβερνοεγκληματικότητας που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Τώρα, όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, χρειάζεται συγκεκριμένη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα όσον αφορά τι αποστολέ αυτού του οργανισμού και σε επίπεδο βιομηχανικό πρέπει να προωθηθεί ενεργά, πολύ ενεργά, ο τομέα τη κυβερνοασφάλεια και του CIS, του Ευρωπαϊκού Συστήματο ε, Πληροφοριών, και όλα αυτά στα πει των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής ε, Task Force για την άμυνα. Προτείνουμε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία αποτελούν συστάσεις που θεωρούμε ότι μπορεί να τα καταλαβαίνει ε, ο πολίτης και που δείχνει ότι υπάρχει βούληση στην Ευρώπη να προαχθεί η άμυνα και η ασφάλεια. Όσον αφορά τα παραδείγματα της Βαϊμάρης, της Βαϊμάρης ΣΥΝ ή της συνεργασίας ε, σκανδινικών χωρών με τη Βαλτική, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν μόνιμες συνεργασίες πλέον, δομημένες και οι συνεργασίε οι διμερεί να χαρακτηρίζονται πλέον ευρωπαϊκέ, παρόλο που είναι πάρα πολύ χρήσιμε. Ε, δεύτερον, θα πρέπει η άμυνα αυτή να πρέπει να έχει την ανάλογη χρηματοδότηση, θα πρέπει να γίνονται προσπάθειε καλύτερη κατανομή των κονδυλίων, 20% από ό,τι θυμάμαι αφορούν τον εξοπλισμό. Ε, πολύ χαμηλό ποσοστό. Ε, τρίτο σημείο, πρέπει να ιδρυθεί και να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία που θα έχει καλέ επιδόσεις, που θα βασίζεται πλήρω στα εφιστάμενα εργαλεία. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα προπολογισμό που θα επιτρέπει να εκπληρώνει τι αποστολέ βάσει των τεσσάρων πυλών που αναφέραμε. Χρειάζεται διάλογο όσον αφορά τι πρωτοβουλίε που αναπτύσσονται ε, άλλων φορέων. Θα πρέπει να υπάρχει επιμερισμό των προσπαθείων μέσω pooling και sharing. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπημένη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, κυρίω όσον αφορά την έλλειψη δυναμικού. Ε, κάτι που απεδείχθη στι πρόσφατε αποστολέ και επιχειρήσει θα πρέπει να είναι διτής προσέγγισης, πολιτικοστατιωτικέ οι προσπάθειε. και θα πρέπει να αφορούν την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια οι διτέ προσπάθειε. Τέταρτη πρόταση έχει σαν στόχο τον εντοπισμό, το συστηματικό των προγραμμάτων δράση που μπορεί να είναι κοινά όταν οι μονομένε πρωτοβουλίε δεν είναι δυνατέ έναντι των μέσων που υπάρχουν και των διακυβευμάτων. Τρομοκρατία, κυβερνοεγκληματικότητα, συγκρούσει απόμακρε κλπ. σε μακρινέ περιοχέ του κόσμου. Μετά πρέπει να δημιουργηθεί ένα κέντρο σχεδιασμού και μόνιμη διεξαγωγή επιχειρήσεων Ευρωπαϊκή Ενώσεω κάτι που αντιμετώπισε δυσκολίε κατά το παρελθόν, η διεθνή κατάσταση δεν μα ε, μας οδηγεί στο ότι πρέπει να βρούμε μόνιμε λύσει από αυτέ που με εμπειρικό τρόπο ε, κατεπηγόντω δημιουργήθηκαν κυρίω όταν το ΝΑΤΟ δεν μπορεί ή δεν θέλει να δεσμευτεί και να καταβάλει προσπάθειε όταν αυτό χρειάζεται. Έκτη προσπάθεια θα πρέπει επίσημα το, του, το στρατηγείο του Ευρωπαϊκού Σώματο να ενταχθεί στην ΚΕΠΑ. Τα, τα πέντε κράτη-μέλη συνεργάζονται μόνιμα μα αυτό και θα πρέπει το πλαίσιο και θα πρέπει να είναι παράδειγμα. Μετά θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στρατηγικέ επιχειρήσει στι διάφορε ομάδε στρατηγικέ που υπάρχουν και, στην, και στο γαλλογερμανικό στάτευμα που έχει δημιουργηθεί. Το 1989 δημιουργήθηκε αλλά δεν έχει κάνει επιχειρήσεις ακόμα. Και κάτι εξίσου σημαντικό, παρόλο που είναι τελευταίο, συστηματική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση όσον αφορά τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, με εύλητο τρόπο από τους πολίτες, χρειάζεται συνέχεια κοινοποίηση όλων τους πολίτες και έτσι θα δοθεί μια νομι... μεγαλύτερη νομιμότητα στον τομέα, άμα καταλαβαίνουν οι πολίτες. Λοιπόν, όλες αυτές οι προτάσεις έχουν κυρίως επιχειρησιακό χαρακτήρα, αλλά έχουν και πολιτικές στοιχείε και περισσότερο θα, θα αναφερθεί σε αυτή την πτυχή ο πρέσβης ο κύριος Μορέλ. Λοιπόν. Ωραία, με προλάβατε. Παρουσιάστε εσείς τον πρέσβη Μορέλ και κυρίως ε, μας ενδιαφέρουν και οι παρασκευαστικές εργασίες για τη Σύνοδο Κορυφής ε, του Δεκεμβρίου. Και καλωσορίζω και τον ε, δεύτερο πρέσβη, τον κύριο Πίτερ Λίχ. Ο πρέσβης Μορέλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, δέκα χρόνια μετά τη Λευκή Βίβλο για την Ασφάλεια το 2003, που επιβεβαιώθηκε το 2008, είναι και η ώρα να ασχοληθούμε με μια μεθοδική ανάλυση της κατάστασης της ασφάλειας στην Ευρώπη. Γι' αυτό και σας παρουσιάσαμε κάποια θέματα και από θεωρητική αλλά και από πρακτική άποψη. Δεν είναι μόνο μια ακαδημαϊκή νοητική εργασία. Θα σας προτείνω εγώ κάποια βασικά θέματα της ανάλυσης και των προτάσεών μας, προσπαθώντας να είμαι όσο πιο απλός και κατανοητός γίνεται. Καταρχήν έχουμε νέα στοιχεία στο πλανήτη και ο κατακαιρματισμός ε, των ε, ε, διαφόρων παγκοσμίων δυνάμεων έφτασε, έδειξε το τέλος στρατηγικής των δύο πόλων. Ο ψυχρός πόλεμος και η εποχή του ψυχρού πολέμου έχει σταματήσει. Τώρα πια έχουμε διάφορα κέντρα και πόλους εξουσίας ε, που δεν είναι ε, προσδιορισμένα απόλυτα, είναι, ε, δεν είναι στατικά και υπάρχει ένα σύστημα μεταξύ πολυκεντρισμού και αναρχίας αρχίζουν και διαγράφονται κάποιοι πόλοι, αλλά είναι κάπως ευμετάβλητοι, είναι αναδυόμενες δυνάμεις που θέλουν να διεκδικήσουν τη θέση τους, αλλά το σύστημα δεν έχει ακόμη αποκρισταλωθεί. Αντί να περιθωριοποιηθούμε σε αυτή τη σύγχυση, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με τις επιλογές της να προσανατολίσει τις εξελίξεις μιας αβέβαιης προς το παρόν διαδικασίας και με μία, ε, αντί να έχουμε μία ε, οικειοθελώς απεσιόδοξη στάση, θα πρέπει να έχουμε μία πολύ ισορροπημένη προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα, ούτε να θεωρούμε ότι είμαστε πρωτοτελεσμένο γεγονότος. Όχι, το παλιό διπολικό σύστημα που ήταν το κληροδότημα το, της δεκαετίας του 50 και που παρατάθηκε στα πλαίσια της του ψυχρού πολέμου έχει ε, παρέλθει ανεπιστρεπτή. Έχουμε δύο συστήματα εδώ και δύο λογικές. Αφενός της πολυμέρειας, γιατί πριν από δέκα χρόνια ε, ευλόγως ταχθήκαμε υπέρ μιας αποτελεσματικής πολυμέρειας. Τώρα όμως έχουμε μια βεσφαλιακή προσέγγιση, είναι βεσφαλιακή, δύο νέους πόλους, δύο δυνάμει, ε, νέες δυνάμεις που αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να χειριστούν, να διαχειριστούν τις εντάσεις. Και με την ε, ανάδυση νέων ε, δυνάμεων ε, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Είχαμε το παράδειγμα της κρίσης της, Συρίας που, της Συρίας που έδειξε την ανικανότητα ε, ανέβρισης μιας λύσης εξαιτία της ασυμφωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να, να δούμε πώς θα διαρθρώσουμε με πιο μόνιμο τρόπο αυτό το σύστημα. Αναφέρθηκαν τα τεχνολογικά θέματα και οι αδυναμίες και τα κενά που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η ραγδαία εξέλιξη των κοινωνιών που γίνονται όλο και πιο εύθραυστες. Έχουμε μερικά αντιμοντέλα, ριζοσπαστικά κινήματα, πολιτισμικούς και πολιτισμικές και θρησκευτικές αντιπαραθέσεις άνευ προηγουμένου. Επίσης πιο εγωιστικές συμπεριφορές, μεθοδική αφισβήτηση της εξουσίας και γενικώ ε, αντιπαλότητες μεταξύ συστημάτων αξιών και κοινωνικών μοντέλων. Και έχουμε επιπλέον και το περιβάλλον. Βλέπουμε ότι μέσα σε μία δεκαετία η κατάσταση έχει προχωρήσει, αλλά τα μέσα που έχουμε δεν, μπορούμε, δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν. Γι' αυτό διαπιστώνουμε μία συστημική αστάθεια απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που διαβλέπουμε. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει κάποια θέση. Βέβαια είχαμε κλασικές κρίσεις, είχαμε το κόδωνα του κινδύνου στα Βαλκάνια, στον Κάφκασο, στη Λιβύη, στο Σαχέλ. Έχουμε όλο και περισσότερα καμπανάκια που χτυπάνε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις κρίσεις. Επίσης είχαμε την κρίση του ευρώ, της ευρωζώνης, που μπορεί να φαίνεται διαφορετική, αλλά δείχνει τελικά το, το εύρος και την ένταση των κλειδονισμών που μπορεί να πλήξουν το σύστημα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε επίσης ε, ε διάφορες εθνικές αντιπαλότητες στο θέμα του πολλαπλασιασμού των όπλων ε, ή ε, ακραίες μεταναστευτικές ροές. Δεν θέλω να δραματοποιήσω τα πράγματα, αλλά βλέπετε τι παράγοντες αποσταθεροποιητικούς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σε μια ορθολογική στρατηγική ανάλυση. Επίσης, έχουμε και συγκεκριμένες εξαρτήσεις της Ευρώπης, συστήματα μεταφορών, επικοινωνιών, ανεφοδιασμού. Είμαστε πολύ ανοιχτοί στον κόσμο, είμαστε εξαρτημένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή την εξάρτηση θα πρέπει να την συνειδητοποιήσουμε, γιατί μας κάνει πιο ευάλωτους. Δεν είμαστε όμως οι μόνοι ευάλωτοι στον κόσμο. Πώς μπορούμε όμως να προσεγγίσουμε αυτή τη νέα κατάσταση, γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι παράγοντες και είπα νεοβαστιφαλική προσέγγιση, γιατί φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο εφαρμόζουμε τις παλιές συνταγές και οι διεθνείς οργανώσεις που εφαρμόζουν την πολυμέρεια και αυτές ε, εξεγείρονται και φαίνεται ότι προτιμούν μια πιο ε, ε, συντηρητική στάση, εκόντες άκοντες. Οπότε έχουμε μία κατάσταση συγκεκριμένη για να μην πω ένα στρατηγικό κενό. Αυτή η κατάσταση δεν είναι κατά ανάγκη αρνητική για την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα πιο ανοιχτό σύστημα, πιο ανταγωνιστικό, κατά πάσα πιθανότητα και πιο τεταμένο, αλλά μπορεί εκεί να βρει νέα περιθώρια δράσης και μια και οι δεν φαίνεται ότι θέλουν να αναλάβουν το έλεγχο του συστήματος και η εξέλιξη του συστήματος μας ενδιαφέρει. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να προλάβει τα πράγματα και να δεσμευτεί, να εμπλακεί σε αυτά. Νομίζω ότι είναι πολύ ρεαλιστική αυτή τη θέση. Και μετά την κρίση τον Κάφκασο ή τις αντιπαραθέσεις στην Κεντρική Ασία, πιστεύουμε ότι η Ευρώπη χωρίς πολυθόρυβο με άμεση αντίδραση να προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις. Γιατί αν ε, κάνουμε μια πιο γενική ανάλυση λιφάνια, θα έχουμε μια θα καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις αντί να αποθαρρυνόμαστε και να, να μπλοκάρουμε μόνοι μας τη λύση. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μια πολιτική και εμπορική ε, δύναμη και θέλουμε, προσβλέπουμε στο να γίνουμε και μια πολιτική δύναμη. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει όμως προσπάθειες και δέσμευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα, θα θυσιάσουμε τις αξίες μας, την ταυτότητά μας, το σήμα κατά τεθέν μας κατά κάποιο τρόπο. Απλώς θα προσδιορίσουμε καλύτερα, θα διαμορφώσουμε καλύτερα αυτή τη στρατηγική που εμείς σας και αγραφήσαμε με αδρές γραμμές. Ο καθηγητής Εμινατόρε μίλησε για την σκληρή στρατηγική, πολιτική, οικονομική, ε, ελαστική απέναντι στους γείτονες, αλλά και πολιτιστική, γιατί τις ε, αρχές και τις αξίες της, προσπαθεί να τις μεταλαμπαδεύσει και προς τα έξω. Πιστεύω ότι σε όλα αυτά θα έχουμε ένα κοινό εγχείρημα με συνοχή. Τώρα, σε γεωπολιτικό επίπεδο, ποια μπορεί να είναι η προσέγγιση μας. Έχουμε εδώ τέσσερα σημαντικά τμήματα, γιατί βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο μεταξύ του, του ευρωατλαντικού χώρου, του ευρωασιατικού χώρου, του ευρωμεσογειακού και αφρικανικού χώρου και ας μην ξεχνούμε και το ευρωαρκτικό χώρο. Να μην ξεχνούμε και αυτή τη διάσταση. Ο ευρωατλαντικός χώρος ε, φυσικά χαρακτηρίζεται από τις, σχέσεις, τις εταιρικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπάρχει μια επανισορρόπηση που είναι ορατή σε όλους. Θα πρέπει να βρούμε ένα νέο τρόπο κατανομής των ευθυνών. Δεν είναι βέβαια μια σημαντική κρίση, δεν είναι εντάσεις αντίστοιχες με αυτές του ψυχρού αλλά έχουμε δύο μεγάλες δυνάμεις που θέλουν να γίνουν παγκόσμιοι ε, παίκτες και θέλουν φυσικά μια έχουν ομοιότητες αλλά έχουν και σημαντικές διαφορές και σε, σε αυτόν τον ευρωατλαντικό χώρο θα πρέπει να λάβουμε και νέες αναδυόμενες δυνάμεις όπως τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική. Ευρωασιατική, ευρωασιατικός τώρα χώρος. Εκεί αποφασιστικό ρόλο έχει η Ρωσία και μπορεί να έχουμε μια πιο σταθερή αρχιτεκτονική και καλύτερα συντονισμένη με τον ευρωπαϊκό χώρο. Άρα θα πρέπει να γίνουν κάποιες επιλογές που δεν έγιναν ούτε από τους μεν ούτε από τους δε ενδιαφέρει την ασφάλεια της Ευρώπης, τη γειτονία της, ενεργειακά ζητήματα, σχέση με την Μέση Ανατολή. Δεν αποκρισταλώθηκαν ακόμη αυτές οι επιλογές. Το ίδιο ισχύει και για την Κίνα, τις Ευρωσιάτες εταίρους και τις αναδυόμενες οικονομίες. Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια διστακτικότητα στο να επιλέξουν την Ευρώπη. η απροθυμία ακόμη. Από τη στιγμή που δεν γίνουν αυτές οι επιλογές και από τους μεν και τους δε, δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις. Μπορεί να έχουμε βλέψει για κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχουμε, βρεθεί ακόμη σε αυτό το, δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το επίπεδο. Και όταν θα συνάψουμε τέτοιες στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, μπορούμε να προσθέσουμε και την πτυχή της ασφάλειας. Βέβαια, πόρο απέχουμε από κάτι τέτοιο, αλλά είναι δρόμος που πρέπει να γίνει. Και μάλιστα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία δεδομένων των κρίσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Εύρω, Εύρο-Μεσογειακό-Αφρικανικός Αφρικανικό χώρο. Σημαντικό χώρο, γιατί κανένα άλλο παγκόσμιο πόλο δεν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την ευρύτερη ζώνη. Και στην ζώνη Μεσογείου Ανατολή ή και στις υποδιαιρέσεις. Έχουμε και ιστορικούς δεσμούς που μπορούμε να τους ε, εκμεταλλευτούμε παρά τις καθυστερήσεις που σημειώσαμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Πρέπει να κινητοποιήσουμε τους πόρους μας και στην Αφρική, γιατί εκεί είμαστε οι μόνοι που προτείνουμε πραγματική συνανάπτυξη. Οι άλλοι προτείνουν κάτι διαφορετικό, όχι όμως ε, ανάπτυξη με ίσους όρους. Ε, νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε στην περιοχή της Αφρικής. Στον Εύρο-Μεσογειακό Αφρικανικό χώρο έχουμε μια διεκδίκηση που την αναγνωρίζουμε, της ε, αξιοπρέπειας, ε, και της, της εθαγένειας και της ε, ασφάλειας. Ε, επίσης, στα πλαίσια της αραβικής και το ενδιαφέρον που δείξαμε για την, Ευρω... για την αραβική άνοιξη είναι ενδεικτικό. Επίσης, ό,τι αφορά τον ευρωακτικό χώρο και για λόγους περιβάλλοντος αλλά και για λόγους στρατηγικής και διάρθρωση των νέων πόλων και ο ευρωακτικός χώρος είναι σημαντικός και άμεσο ενδιαφέρον για μας. Δεδομένων όλων αυτών των συνιστοσών, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις, κάποιο ξεκαθάρισμα με τους εταίρους μας και σε αυτές τις ε, γεωγραφικές ζώνες να κάνουμε και νέες προσπάθειες ή τουλάχιστον να προτείνουμε μια στρατηγική επανακινητοποίηση της Ευρώπης με μια πιο παγκόσμια προσέγγιση. Τώρα η μεταμόρφωση του στρατηγικού πλαισίου μας υποχρεώνει να ασχοληθούμε και με το θέμα της ασφάλειάς μας στις επόμενες δεκαετίες. Και η αποκλειστική επιλογή του Smart Power ε, είναι ε, μόνο ε, φαινομενικά καλή λύση. Γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε τους δυνητικούς αντιπάλους μας να χρησιμοποιήσουν χειραγώγηση ή την ε, ισχύ τους προκειμένου να παρακάμψουν την αποκλειστική μας επιλογή της έξυπνης στρατηγικής. Δεν μπορούμε εμείς να θυσιάσουμε τους άλλους πόλους της δύναμης. Οπότε θα πρέπει φυσικά να επικεντρωθούμε στη δυτική χρήση, στρατηγική και πολιτική, αλλά ε, ας μην αποκλείσουμε και σε περίπτωση ίστα της ανάγκης και σε περίπτωση άμυνας τη χρήση και της ε, στρατιωτικής δύναμης γιατί φυσικά χρειαζόμαστε μία σύγκληση στα θέματα της ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι απαραίτητο θέλουμε να συμβάλλουμε στην οργάνωση του παγκόσμιου συστήματος, δίνοντας τις σωστές απαντήσεις που είναι οι μοναδικές που χρειαζόμαστε δεδομένης της εξέλιξης ε, του παγκόσμιου συστήματος. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Λεωκιός Πρεσβευτής, Φίκος Μπίτερλιχ. Κύριε Προέδρε, κυρία Αντιπροέδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Οι τρεις συνάδελφοί μου παρουσίασαν τέλεια τα ουσιαστικά στοιχεία των εργασιών που διεξήχθησαν εντός του κέντρου στατικών ερευνών στις Βρυξέλλες και αναφέρθηκαν σχεσιμότητα, σκοπιμότητα και αναγκαιότητα η Ευρωπαϊκή Βίβλος, η Λευκή Βίβλος της Άμυνας να υπάρξει ε, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιχειρησιακής φύσεως σε σχέση μάλιστα με αυτά που έγινε το 2003. Βλέποντας πώς έχει προχωρήσει η συζήτηση, θέλω να προσθέσω κάποια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, η αποτίμηση, απολογισμός από Μάστριχτ μέχρι Λισαβόνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να προωθήσει την ιδέα μιας κοινή εξωτερικής πολιτικής και μιας κοινή πολιτικής ασφαλείας. Οι πρόοδοι έκτοτε είναι μικρές, υπάρχει μια, ε, ένας κατάλογος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αρκετά σημαντικός κατάλογος που αυτόματα πάντα αποδεικνύει τα, όρια των δυνατοτήτων μας. Και είναι περιορισμένη η πρόοδος γιατί. Διότι ε, διατηρήσαμε κάποιες, κάποια εθνικά αντανακλαστικά και ήμασταν και περιορισμένοι κάπως λόγω των σχέσεων με τον ΝΑΤΟ. Κυρίες και κύριοι, τα όρια αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο επειδή ο κόσμος γύρω μας άλλαξε ριζικά, αλλά διότι οι στρατοί μας υποχρηματοδοτούνται. Αυτό δεν είναι νέο φαινόμενο, αλλά είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε εδώ και περίπου 20 χρόνια. Χρηματοδότηση, περιπλοκότητα των κρίσεων και των συγκρούσεων και ο κόσμος που αλλάζει γύρω μας αφήνει μόνο μία επιλογή θα πρέπει να υπομισθούμε τις ευθύνες μας και ταυτόχρονα θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, τα μέσα μας, τα εργαλεία μας. Ε, αυτό σημαίνει καταρχάς από την αρχή να ξεκινήσει μια εις βάθος συζήτηση με βάση τα τρία ερωτηματικά. Πρώτα απ' όλα, αξιολόγηση του κόσμου. Δεύτερον, ποιο είναι το όραμά μας στο στατικικό και ποια είναι η θέση μας στον κόσμο. Και τρίτον, δομές, μέσα και εργαλεία. Ομολογώ ότι πάντα υπερασπιζόμουν τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Στατού τελικά. Και πιστεύω ότι έχει οριμάσει η ιδέα, εξού και η ιδέα να προχωρήσουμε προς το αποκαλούμενο pooling and sharing, ένωση δυνάμεων, συνένωση δυνάμεων, αλλά με σοβαρό τρόπο να προχωρήσουμε πραγματικά και να μην μείνουμε στο πρώτο κομμάτι της διαδρομής. Πιστεύω ότι είμαστε στην απαρχή μιας τέτοιας συζητήσης. Αυτή η συζήτηση καμιά φορά ε, προκύπτει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που δεν μπορώ να κρύψω, ακόμα και αν ο φίλος μου Πιέρ Μορέλ είναι δίπλα μου. Τον Ιανουάριο, όταν ξέσπασε η σύγκρουση στο Μαλί, ε, ήμουνα στο Αλγέρι, με είχε προσκαλέσει η κυβέρνηση που μου πρότεινε την ιδέα ότι οι Γάλλοι ε, θα πρέπει να συνοδευτούν από την Ευρώπη να γίνει τουλάχιστον επιχειρήσει υπό την αιγίδα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Γιατί? ούτω ώστε να υπάρχει καλύτερη προστασία των Γάλλων στην Αφρική. Εγώ θεώρησα ότι ήταν έξοχη η ιδέα αυτή. Γνωρίζω ότι ακόμα και οι διαδικασίες οι υπάρχουν, αλλά ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν. Καταλαβαίνω ξαφνικά βέβαια από την άλλη πλευρά ότι η Γαλλία προτίμησε λόγω των περιστάσεων να δράσει γρήγορα. Και οι ίδιοι και οι Αλγερινοί το κατάλαβαν αλλά εγώ κάπου αισθάνθηκα θλίψη, διότι αυτή η επιχείρηση δεν μπόρεσε να λάβει χώρα υπό μια ευρωπαϊκή σημαία. Ε, Κυρίε και κύριοι, κάποιες πρακτικής φύσεως ε, που θα έπρεπε ή θα μπορούσαν να τεθούν πριν ή και στην αρχή των εργασιών ε, για την επεξεργασία μιας διευκής βίβλου ευρωπαϊκής. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος ε, τρόπος ε, συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν επιφυλάξει σχετικά με αυτό. Ας είμαστε πραγματιστές. Ας προσπαθήσουμε όμως να δημιουργήσουμε ένα είδος μόνιμης συνεργασίας σε αυτό το τομέα για να υπερκεράσουμε τις διαφορές, τις επιφυλάξεις και να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ αυτών των φορέων νομιμότητας. Δεύτερον, διαθέτουμε κάποιες αρχές δομών, απαρχές δομών ευρωπαϊκής φύσης εδώ στις Βρυξέλλες και στο Συμβούλιο, αλλά διαθέτουμε πάνω απ' όλα την, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, που θα έπρεπε να οικοδομηθεί σαν μια ευρωπαϊκή κεντρική υπηρεσία. Θα πρέπει ε, γρήγορα να ε, οδηγηθούμε σε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά την, τον εφοδιασμό, τους διαγωνισμούς για τους εξοπλισμούς μέσω αυτού του φορέα και θα πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα να γίνει συντονιστικό φορέα τη έρευνα που απαιτείται και τη ανταλλαγή υλικού, αμυντικού υλικού που απαιτείται. Τρίτη ιδέα, πολύ γρήγορα ρίχνω τι ιδέε. Δημιουργήσαμε τι ομάδε κρούση, μάχη, battle groups. Οι παλιοί στρατιωτικοί μου λένε ότι πρέπει να αντικατασταθούν από κάποια τάγματα ε, για να πρέπει να γίνει πιο εύκολο αυτό το, η χρήση του μέσου αυτού. Ε, μετά από μακρύς δισταγμούς ε, δημιουργήσαμε κάποια ομαδοποίηση των μεταφορικών μέσων, pooling, και που συμπεριλαμβάνει και όλες τις δυνάμεις μας σε ελικόπτερα. Και αυτό είναι πολύ καλή ιδέα, διότι έχουμε δυναμίσει να αφορά τις μεταφορές δεν θα αναφερθώ στη γαλλογερμανική συνεργασία ή την ενισχυμένη συνεργασία διότι, ε, και στο ε, γαλλογερμανικό σώμα, διότι αυτά εξυπακούνται, είναι αυτονόητα. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι οι συνεισφορέ σας, οι παρουσιάσεις προφορικές αυτές δείχνουν τον πλούτο των εργασιών, του γραπτού, της γραπτής πρότασης που έχουμε στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις παρουσιάσεις. Ήταν πολύ ποιοτικέ. Κάποιοι συνάδελφοι ήθελαν να πάρουν το λόγο. Αν είχετε την καλοσύνη, συγχωρήστε με. Ε, έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας, πρέπει να αποχωρήσω. Ε, είμαι πολύ ευτυχής που μπόρεσα να ακούσω όλες τις παρουσιάσεις σας, διότι πραγματικά ήταν πολύ ποιοτικέ. Η Αντιπρόεδρος ε, και Σοφοκλέο θα με αντικαταστήσει. Ο κ. Σοφοκλέο. Ε, και η κυρία Νικολάη θέλει να μας ε, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω τα ρουμανικά διότι η ποιότητα ε, των παρουσιάσεων σας με υποχρεώνει να πω ότι τα γαλλικά μου και τα αγγλικά μου ίσως είναι κάπως φτωχά για να τα αποκριθούν και σε αυτά που θα πρέπει να πω. Χαιρετίζω λοιπόν και εγώ αυτή τη συζήτηση για πρώτη φορά κατά την άποψή μου ήταν μια πολύ ε, προχωρημένη συζήτηση, μια προσέγγιση ε, που από το 1989 πιστεύαμε ότι είναι χαρακτηριστική για την Ανατολική Ευρώπη. Και συνέβαλε εν μέρη στην πτώση του ε, κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε κάποια έγγραφα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διατύπωση μπλοκάριζε την ιδέα και το όραμα και προφανώς και, την, και τις αποφάσεις. Στη σελίδα 65 του εγγράφου στρατηγική για την ασφάλεια, εκεί προτείνεται ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ε, μια ευρωπαϊκή λευκή βίβλος και πολλοί από εμάς μήπως ε, αυτό είναι ένας δούριος ε, ύπος ο οποίος κατά κάποιον τρόπο θα καθυστερήσει τη λήψη αποφάσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, και πρέπει να διερωτηθούμε κατά πόσον ε, χρειαζόμαστε ένα όραμα στον τομέα της ε, ΚΕΠΑ και κατά πόσον γνωρίζουμε πού ακριβώς θα βρισκόμαστε τα επόμενα 20 ή 30 χρόνια. Ο κύριος Μορέλ μίλησε για την έλλειψη οράματος. Βεβαίω, αν η στρατηγική 2020, η οποία ξεκίνησε από τον Deng Xiaoping, μετά από τον Medvedev και μετά ε, συνεχίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αυτό είναι όραμα, εμείς ε, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει όραμα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε ε, ότι εκείνο που ε, μας δίνει ένα όραμα είναι η πολυπολικότητα. Σήμερα ζούμε σε ένα κόσμο με ένα και πόλο, της Ηνωμένε Πολιτείε. Αν όμως δούμε λιγάκι γύρω μας, προφανώς ε, η λύση έγκυται στην πολυπολικότητα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επανέλθω σε θέματα ε, πολιτικών ασφαλείας. Εγώ πιστεύω ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να την επανεφεύρουμε με, με λίγα μονοθέματα και η ΚΕΠΑ είναι ένα από αυτά. Αυτό λοιπόν σημαίνει τεχνολογική και βιομηχανική βάση που θα είναι κοινή για όλους μας και αυτό θα επιτρέψει την επανεφεύρεση της Ένωσης. Γιατί αν δούμε ψύχρεμα τα προϊόντα που μπορούμε να παράγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταλήξουμε στο ότι τα ευρωπαϊκά αεροσκάφη είναι πολύ γνωστά ανά τον κόσμο. Άρα δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είμαστε ανταγωνιστικοί σε τομέας που έχουμε παράδοση και ποιότητα και αυτό λοιπόν αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για μας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια λευκή βίβλωση για την ασφάλεια, αλλά κάτω από μια προϋπόθεση. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα μέσο μακροπρόθεσμο όραμα, ε, θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να κατανοήσουν ότι όλοι οι κίνδυνοι για επικυριαρχία μπορούν να καταστρέψουν αυτή την περιοχή. Και αν υπάρξει καταστροφή, αυτομάτως ε, θα υπάρξει και κατακαιρματισμός. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τη σημασία μας στο γεωπολιτικό παιχνίδι βραχυπρόθεσμα και μέσοπρόθεσμα. Άρα δηλαδή αυτά που δεν έχουν σχέση με την πολιτική είναι απαραίτητο να εξεταστούν. Δυστυχώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν όραμα και αυτό κατά την άποψή μου είναι ένας από τους λόγους που δεν προχωράμε προς τα εμπρός. Αυτό ελέγχθη κάποτε και στο πλαίσιο του συνεδρίου στο Παρίσι. Πρέπει λοιπόν να ε, δημιουργήσουμε ένα όραμα που θα ιεραρχεί τους ε, κινδύνους. Ας δούμε ποιοι είναι οι κινδύνοι με τους οποίους θα έρθουμε αντιμέτωποι τα επόμενη 20-30 χρόνια. Από στρατηγική σκοπιά πιστεύω ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τοπικούς ε, πολέμους, τοπικής εμβέλειας, όπου ο Ευρωπαϊκός στρατός μπορεί να είναι χρήσιμος για τη διαφύλαξη της ειρήνης και για την επαναφορά της τάξης. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό στρατό, γιατί αυτό είναι πιο φτηνό, μας καθιστά περισσότερο σύμβατους τον ένα με τον άλλο ε, και επίσης ε, ε, υπάρχει αλληλένδεση ανάμεσα στους διάφορους τομείς και με τον τρόπο αυτό αποδίδεται και διαφορετική σημασία στον, στην έννοια της ε, δύναμης. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ε, συγκεκριμένα μέτρα που προτάθηκαν και εγώ συμφωνώ με αυτά που προτάθηκαν κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος ελευθεριών και δικαιωμάτων και Τώρα όμως φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ε, προστατευτεί ε, να προστατεύσει τις ελευθερίες της και τα δικαιώματά της. Αυτές λοιπόν οι ελευθερίες βοήθησαν να ε, διαφυλαχθούν κάποιες αξίες και από ό,τι φαίνεται πόσο ευάλωτοι είμαστε όταν πρόκειται για την προστασία των συμπερόντων των Ευρωπαίων πολιτών η ικανότητά μας ε, να αντιδράσουμε πρέπει να είναι προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να υπάρχει μια επικοδομητική συνεργασία με τα κράτη-μέλη γιατί με τον τρόπο αυτό η αντιδράση μας ε, μπορεί να είναι διτής φύσεως. Όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών, εκεί εγώ έχω λιγάκι διαφορετική άποψη. Εμείς πιστεύουμε ότι στον τομέα αυτό υπάρχει ανταγωνισμός. Βεβαίως υπάρχουν εδώ κάποιες πολιτιστικές αξίες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε τις, τους πόρους, να τους καταστήσουμε συμβατούς μεταξύ τους, αλλά ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τον ανταγωνισμό. Δεν πρέπει να δούμε τα θέματα όπως τα βλέπουν οι Γερμανοί. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε ε, χωρίς ε, βέβαια να περιζόμαστε μόνο στα πολιτιστικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε διάφορους ε, τομείς. Και πιστεύω επίσης ότι έχουμε εδώ δύο ε, βασικές προτεραιότητες. Τη Μεσόγειο, όπου είμαστε ε, σημαντικοί αλλά και ευάλωτοι και την Ανατολική πλευρά, τον Κάφκασο και την Κεντρική Ασία. Εκεί μπορεί, να, μπορούμε να επιτύχουμε κάποια σταθερότητα και μπορούμε να αποφύγουμε ε, κάτι που μας έχει προσφέρει η ιστορία. Πάντως, αυτά μπορούν να αποτελούν και πηγή συνεργασία στον οικονομικό τομέα ε, και ε, συνεργασία σε στρατηγικής φύσεως εξαγωγές. Τελειώνοντας, ε, θα ήθελα να πω ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και πιστεύω ότι τελικά μπορεί και να τα καταφέρουμε. Και θέλω να σας πω αυτά που με εντυπωσίασαν. Αυτά δεν ήταν ε, απαραίτητα η συνεργασία για αυτά που είπατε για την Κεντρική Ασία αυτή είναι μια περιοχή που τη θεωρούμε πολύ σημαντική. Αυτό που μας εντυπωσίασε είναι το γεγονός ότι εμείς μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους, από τους Αμερικανούς, τους Ασιάτες, τους Κινέζους, γιατί έχουμε και τη δυνατότητα να σκεπτόμαστε διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν εφόσον μας προσφέρεται μια ευκαιρία, είναι κρίμα να μην τη χρησιμοποιήσουμε πολιτικά και είναι κρίμα να μην υπάρχει λευκή δίπλωση ε, για την ασφάλεια. Μπορούμε να τη συντάξουμε πολύ γρήγορα, μπορούμε να επηρεάσουμε τις αποφάσεις και αυτό μπορεί να δώσει και την ευκαιρία να επανεφεύρουμε την Ευρώπη. Κρόνμπερκ έχει Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που μας είπε ο καθηγητής Σεμινατόρε για την ε, στρατηγική ασφάλειας, την ενιαία στρατηγική ασφάλεια. Συμφωνώ ότι η Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μία ενιαία στρατηγική ασφάλειας και όχι 27 και σύντομα 28 διαφορετικές. Βέβαια θα πρέπει για να έχουμε κοινή στρατηγική ασφάλειας να έχουμε μία κοινή αντίληψη των απειλών που υπάρχουν. Και εκεί είναι που έχουμε κάποια κενά. Στην υποεπιτροπή μας εξετάσαμε την πιθανότητα ε, να δούμε τις απειλές που αντιμετωπίζουν ε, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ευρωπαϊκά έθνη. Αλλά δεν καταφέραμε τελικά ε, να το συζητήσουμε. Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια κοινή αντίληψη περί απειλής ή τουλάχιστον διαφορετικές αντιλήψεις για απειλές. Η στρατηγική του 2013 μιλούν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία και τις ε, χώρες που χαρακτηρίζονται από αναρχία. Έχουμε ένα τέτοιο ε, κράτος πολύ κοντά σε εμά, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε μια στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να το αντιμετωπίσουμε. Ε, μία από τις κοινέ απειλέ θα μπορούσε να είναι η διάδοση των πυρηνικών όπλων. Εξαιτία τη εύκολη πρόσβαση στην πυρηνική τεχνολογία, Βόρεια Κορέα, Ιράν, δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα και ίσω στο μέλλον θα αποκτήσουν πρόσβαση και άλλες χώρες. Είχαμε την Ορβηγική Διάσκεψη για τις ανθρωπιστικές συνέπειες ε, ενός μικρού, μικρής εμβέλειας πυρηνικού πολέμου. Και το συμπέρασμα ήταν ότι καμία χώρα στον κόσμο θα μπορέσει να διαφυλάξει τους πολίτες της από μία πυρηνική έκρηξη, από μία έστω και μικρής εμβέλειας πυρηνική σύγκρουση. Έχουμε και και εσωτερικές απειλές στην Ευρώπη. Το χάσμα μεταξύ πλουσίου και φτωχών που όλο και διευρύνεται και που εξωθεί στην περιθωριοποίηση ορισμένων στρωμάτων και δημάτων του πληθυσμού, κάτι που δημιουργεί μια κοινωνική αναταραχή. Για να κοιτάξουμε την κατάσταση στην Ευρώπη με μια ευρύτερη προοπτική και δεκαετή, ίσως και εικοσέτη. Ερωτώ λοιπόν, με ποια διαδικασία θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει μία νέα αντίληψη για το ποιες θα είναι στο μέλλον οι απειλές που θα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φοβάμαι ότι διαφωνώ κάθετα με την κατεύθυνση που ακολουθεί η Λευκή Βίβλος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Νομίζω ότι άμυνα θα πρέπει να σε αρμοδιότητες του ΝΑΤΟ και των κρατών μελών. Το ΝΑΤΟ λειτουργήσε πολύ καλύτερα παρά οποιαδήποτε συνεργασία στα τευμά της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Διαφωνώ με το όλο πνεύμα της τοποθέτησής σας, της μελέτης σας. Κανονικά αυτό είναι ο ρόλος μου, το ξέρω. Αλλά έχω ερώτηση. Κύριε Μπίτερλιτς, ε, προδόθηκε ή αναφέρθηκε σε στρατό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην ίδια αίθουσα του Κοινοβουλίου, στον Ολομένιο του Κοινοβουλίου, το αρνήθηκαν. Δεν μου αρέσει να μου λένε ψέματα, βαρέθηκα. Εσεί εδώ, οι τέσσερι σχολιαστέ, ο καθένα από εσά, πείτε μου ξεχωριστά, θέλετε να υπάρχει ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό στρατό και ενιαία πολιτική ε, ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστέ ειλικρινεί. Διότι αυτό το πείσμα όσον αφορά την πραγματική κατεύθυνση των αμυντικών εγγράφων πρέπει να ξεκαθαριστεί. Εστέ ειλικρινείς αποκαλυφθείτε. Αν θέλετε έναν ενίο στρατό, πείτε το. Και αν θέλετε πολιτική ένωση, πείτε το. Διότι νομίζω είναι πάρα πολύ επικίνδυνο έδαφος αυτό. Και κάτι άλλο ερώτημα. Η δικαιολογία στις επιτροπές αυτές είναι ότι πάντα υπάρχει υποχρηματοδότηση. Το είπατε κι εσείς. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μία ε, δικαιολογία για να συλλέξετε δυνάμεις για να προωθήσετε τον πολιτικό σας σκοπό. Και εσείς οι τέσσερις κύριοι Πείτε μας, υπάρχει πρόγραμμα κρυφό να ενωθούν οι άμυνες, να καταργηθούν μάλλον οι άμυνες σε επίπεδο κρατών μελών για να δημιουργήσετε αυτό τον Ευρωπαϊκό Στρατό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εστέ ειλικρινείς, έχω βαρεθεί με τα ψέματα που ακούσα αυτή την Επιτροπή. Τα άκουσα επανειλημμένα, είμαστε ειλικρινείς. Ας ακούσουμε το πραγματικό πρόγραμμα για αυτή την άμυνα. Σας ευχαριστώ. Πολλά ερωτήματα και τώρα είναι η ώρα των απαντήσεων. Θα δοθεί ο χρόνος στους φιλοξενούμενους μας ξεκινώντας από τα αριστερά μου όπως καθόμαστε να δοθούν οι απαντήσεις οι σχετικές. Je me... Je me limiterai Θα περιοριστώ σε μία απόπειρα απάντηση στην κυρία Βουλευτή. Πρέπει να πω ότι βάσισα την όλη μελέτη μου επί του Διεθνούς Συστήματος της Διπολικότητας και το έκανα αυτό με τη συνεργασία επιφανών προσωπικότητων της γαλλικής στρατιωτικής θεωρίας. Τότε που υπήρχε το αποτρεπτικό, το διπολικό, το deterrent, η αποτρεπτική πολιτική και η στρατηγική της ε, ελάχιστης προσπαθίας η γαλλική, της μικρής προσπάθειας. Και διαταράκτης είχε την έννοια το να επιδεινώσει κανείς κάθε κίνδυνο για πυρηνική σύραξη που θα οδηγούσε σε μια γενοκτονία. Η σημασία του πυρηνικού όπλου όπως την ε, διδάχτηκα είτε είναι διπολική ή πολυπολική ποια είναι. Να καθορίσουμε το πυρηνικό όπλο σαν ένα όπλο που δεν χρησιμοποιείται. Ε, μελετήσαμε τότε τις ενδεχόμενες συνέπειες πυρηνικής σύραξης, περιορισμένου πυρηνικού πολέμου, μικρής κλίμακας. Συμφωνούμε μελέτη της Νορβηγίας ότι η περιορισμένη πυρηνική σύγκρουση που προβλεπόταν στο κεντρικό μέτωπο τότε θα ήταν κάτι καταστροφικό και θα εμπόδιζε ακόμα και, τους, ε, και τις κινήσεις και τους ολιγμούς των μεγάλων μονάδων. Ε, θυμάμαι τη βίβλο της Σοβιετικής Άμυνας τότε που λεγόταν «Επίθεση» ήταν ο τίτλος της. Ξεκινούσε λέγοντας στα πλαίσια μιας γενικής στρατηγικής αμυντικής, η, Σοβιετική Ένωση, ζητώ συγγνώμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη που είπα αυτό, δίνει εντολή στο στρατό να ξεκινήσει μια σύγκρουση με όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων και των πυρηνικών μέσων. Αυτό θα ήταν αδύνατος ελιγμός για τους στρατούς του Συμφώνου της Βαρσοβίας στο κεντρικό μέτωπο και αδυναμία ακόμα να μελετηθεί τον δεχόμενο περιορισμένου πυρηνικού πολέμου. Δεν υπάρχουν παραδείγματα επί των οποίων να βασιστούμε. Η σημασία του πυρηνικού όπλου μέχρι τώρα ε, ήταν η διπλωματική χρήση. Και τότε την εποχή της διπολικότητας οι συγκρούσεις που εμελετούντο ήταν περιφερειακής φύσεως ή παρεπόμενες συγκρούσεις διότι οι χώρες χρειάζονται απάντηση, να δώσουν απάντηση στη βία προφανώς μέσω μιας βίας που ρυθμίζει την ε, διεθνή τάξη. Ε, το μόνο ερώτημα που τίθεται και αυτό που υπονοείται στην όλη λογική που ακολουθείτε, αυτού που κάνει την ανάλυση του φαινομένου της διάδοσης των πυρηνικών όπλων, είναι το εξής. Οι δυνάμεις που θέλουν να έχουν πυρηνικό όπλο θέλουν να απομονωθούν. Και όταν υπάρχει συνέχεια στατιωτική μεταξύ συμβατικής άμυνας και πυρηνικής άμυνας, η συμβατική άμυνα έχει την ελευθερία δράση που απαγορεύεται στην πυρηνική άμυνα. Αυτό σημαίνει ότι στα πλαίσια του Ιράν, παράδειγμα, αν το Ιράν απομονωνόταν θα μπορούσε πάντα να χρησιμοποιήσει τον πολιτικό του ρόλο και την πολιτική επιρροή και τη στατιωτική σε όλη την περιοχή. Από τον κόλπο μέχρι Κεντρική Ασία μέσω συμβατικών όπλων. Ιδού λοιπόν ποιε είναι οι πολιτικοστατητικέ πτυχέ του πυρηνικού όπλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πυρηνικό όπλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, από του τρομοκράτε, στο τρομοκρατικό επίπεδο. Σε επίπεδο τρομοκρατίας δεν έχουμε προφανώς τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ποια θα ήταν η καταστροφή. Δεν θέλω να δώσω παραδείγματα για να μην τρομάξω εδώ το ακροατήριο, αλλά ας πούμε ένα πυρηνικό όπλο ακόμα και σε πολύ μικρό μέγεθο, σε μια μεγάλη πόλη, μεγαλόπολη, θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα και δεν θα ήταν μόνο αυτό. Προ, σας προειδοποιώ ότι η χρήση από τρομοκράτη ποινικού όπλου πίσω από αυτό υπάρχει υποστήριξη κράτους συνοδεύεται από μια αλυσιδωτή αλληλοχία ε, γεγονότων και δεν θέλω να σας δώσω περισσότερα στοιχεία είναι η μόνη απάντηση που μπορώ να σας δώσω τώρα κυρία μου. Εγώ θα απαντήσω στις ερωτήσεις που θεωρώ ότι μου απευθύνθηκαν. Κύριε Νικολάη, για την πρόταση για μια ευρωπαϊκή υπηρεσία, κεντρική υπηρεσία πληροφοριών. Ε, δεν είμαι αφελής. Γνωρίζω ότι ε, η υπηρεσία πληροφοριών συνήθως είναι εθνικό ζήτημα. Ε, κάποιος που μπορεί κάτι περισσότερο μπορεί και κάτι λιγότερο. Οπότε θα πρέπει πρώτα να έχουμε ένα συντονισμό των πληροφοριών και φυσικά μέσα για να είμαστε αποτελεσματικοί. Μια στιγμή μάλιστα που υπάρχει επικάλυψη μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Τα όρια μεταξύ των δύο είναι πολύ ρευστά και σχεδόν απροσδιορίστα σε μερικές περιπτώσεις. Δεν είμαι ουτοπιστής λοιπόν, ούτε πλήρως εθεροβάμων, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα πρόοδου και στο θέμα αυτό. Τώρα να απαντήσω στον κύριο Κάμπελ για το κατά πόσο είναι χρήσιμη ή όχι μια λευκή βίβλος. Και έχουμε και το θέμα του ΝΑΤΟ. Αν είδατε την, το βιογραφικό μου, θα είδατε ποιο ήταν και το παρελθόν μου και στη διαδρομή του. Ε, ούτως ή άλλω δεν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΝΑΤΟ δεν δικαιούται να έχει επιχειρήσει σε ορισμένε περιοχέ και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί κάλλιστα να συμβάλλει. Και μάλιστα Βερολίνο συν έχει κολλήσει αυτή τη στιγμή για τους γνωστούς λόγους. Και η μόνη αποστολή που έχουμε στα πλαίσια του Βερολίνου ΣΥΝ είναι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Που με το ζόρι συνεχίζεται και μένει σε ζωή. Αλλά με βάση το Βερολίνο ΣΥΝ δεν βλέπω μεγάλες ελπίδες ακόμη. Πάντως θα μπορούσαμε και να σημειώσουμε κάποιο πρόοδο, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμη. Γι' αυτό και είπαμε λευκή βίβλος για να λάβουμε υπόψη της ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πιθανής παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, Ευρωπαϊκός στρατός. Δεδομένου του παρελθόντος και της πείρας μου, Νομίζω ότι θα πρέπει, αν τον αποφασίσουμε τον Ευρωπαϊκό Στρατό, να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Μπορεί να είναι απότερο σκοπός, όχι βραχυπρόθεσμος. Έχουμε όμως κάποια μέσα και μηχανισμούς ήδη που υπάρχουν και που είναι αρκετά δαπανηροί. Και η δυσκολία που έχουμε απέναντι στους συμπολίτε μας, σοβού της κρίση, είναι να τους πείσουμε για ορισμένε αποφάσει ενώ τα κονδύλια που έχουμε επενδύσει ε, σε ορισμένα πράγματα δεν αξιοποιούνται, όπως ε, η γαλλογερμανική μεραρχία ή τα battle groups, αυτές οι μάχημες ομάδες, ε, μονάδες. Είναι υπάρχοντες μηχανισμοί που υπάρχουν και θα μπορούσαν να προβληθούν πολύ περισσότερο, ιδιαίτερα στα πλαίσια των μηχανισμών ε, της ΚΕΠΑ. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά που ήδη υπάρχουν ως ένα πρώτο βήμα. Τώρα για πολιτική ένωση για την πολιτική ένωση. Το μόνο που έχω να πω είναι αυτό που έχουν πει ήδη οι πολιτικοί. Δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα. Σε ό,τι αφορά την υποχρηματοδότηση ως, ε, ε, ή ως πρόσχημα, ε, εγώ είμαι είμαι στρατιωτικό. Οπότε τη στιγμή που μου αναθέτει κάποιο μια αποστολή, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να την υλοποιήσω. Αν δεν έχω τα μέσα όμω να το κάνω, είναι δύσκολο. 30,5 εκατομμύρια της αμυντικής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και τα περισσότερα, ένα μεγάλο τμήμα αφορά διοικητικές δαπάνες και έχει τεράστιες αρμοδιότητες και πάρα πολλές υποχρεώσεις και καθήκοντα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και γνωρίζουμε ότι όλα, όλες οι επιμέρους αρμοδιότητες είναι ε, τεράστιες και ταπανήρες και με, τι να κάνει με 30 εκατομμύρια που είναι ε, περίπου όσο προπολογιζόμαστε του EMTM, που είναι 24 εκατομμύρια. Τι να πρωτοκάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Οπότε όταν ε, έχουμε πολλές φιλοδοξίες θα πρέπει να έχουμε και αντίστοιχα μέσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μεγαλομανείς και ότι θέλουμε να κατασπαταλήσουμε τα κονδύλια των, ε, των Ευρωπαίων πολιτών και φορολογουμένων, αλλά από τη στιγμή που έχουμε κάποιες αποστολές και υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί σε ανώτατο επίπεδο θα πρέπει να προβλέψουμε και τα κατάλληλα κονδύλια. Κύριε Κάμπελ, παίρνετε το στατηγικό ρόλο του διαταράκτη και αυτό με χαροποιεί. Αλλά δεν αποκαλύψετε τις προθέσεις σας. Απλώς δώσατε ριζοσπαστική, δώσατε φύση στις απόψεις των άλλων. Δεν προτείνατε εσείς κάτι. Ποια είναι η δική σας πρόκληση. Έχετε κάποιες ιδέες να προτείνετε. Αυτό που προτείνουμε, αφήστε με τελειώσω, αυτό που προτείνουμε είναι ένα μέσο, εργαλείο γενικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, σταδιακά και διαφοροποιημένα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολιτικά. Παράδειγμα, ενώπιον της Συρίας που είναι η πρώτη πολυπολική σύγκρουση, η Μεγάλη Βρετανία έχει ένα όραμα. Η Λευκή Βίβλος σημαίνει να έχουμε ένα όραμα εντός του οποίου να δράσουμε και τα μέσα δράσης και οι στόχοι ίσως σταδιακά να καθορίζονται. Σήμερα η Μεγάλη Βρετανία έχει ένα όραμα για τη Συρία και αυτά που πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ κύριε Κάμπελ. Ε, απάντησε κύριος Μορέλ. Ε, κύριος Μορέλ έχει τον λόγο. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Θα απαντήσω πρώτα απ' όλα στην κυρία Νικολάη όσον αφορά τα σχόλια και τις αναφορές τις γαλλικές στη Λευκή Βίβλο. Θα πρέπει να τα δει κανείς θετικά. Ε, τα βλέπω ανεξάρτητα τα πράγματα. Δεν εξυπηρετώ πλέον τους σκοπούς της ε, γαλλικής δημοκρατίας. Είμαι ανεξάρτητος πολίτης. Είναι αξιοσημείωτη αυτή η Λευκή Βίβλος για την άμυνα σε μια περίοδο πολύ δύσκολη λόγω, για λόγους οικονομικούς. Ε, αντιστοιχεί σε έξι ε, μήνες μεγάλων πνευματικών προσπαθειών, ποιοτικών. Αυτό πρέπει να το γνωρίσουμε και υπογραμμίζει την ανάγκη της Ένωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, βλέπω ένα μήνυμα, μία έκκληση από πλευράς μιας λογικής στα πλαίσια της γαλλικής παράδοσης. Δηλαδή, η Γαλλία πρώτη κανονικά, η Γαλλία έχει προτεραιότητα, είναι η γαλλική προσέγγιση. Βέβαια πρέπει να γίνονται εθνικές επιλογές, αλλά στο τέλος, στο κάτω-κάτω της γραφής, η ε, υπάρχουν κάποιες επιλογές που πρέπει να γίνουν οικονομικές και πρέπει να αναγνωριστεί ότι είναι απαραίτητη ε, μια ιστορική συμπληρωματικότητα που επιβάλλεται. Ε, στα 40 χρόνια κινούμε στον χώρο της ασφαλείας της Γαλλίας. Θεωρώ ότι αν ακόμα δεν αναφέρεται με μεγάλα λόγια, αν διαβάσετε προσεκτικά το έγγραφο, θα διαπιστώνετε ότι είναι σημαντικός, σημαντικός κόμβος διανοητικός, θεωρητικός για τη συνέχεια. Δεν προδικάζει τίποτα παρατείνει αν θέλετε, ε, επεκτείνει αυτό που αναφέρθηκε στην έκθεση Βεντρίν όσον αφορά την Ατλαντική Συμμαχία ε, με τον Κιμπέρ Βεντρίν είδα τι συνομιλίες που έγιναν ε, το αναγνώριζε ότι δεν, καλε, δεν εκαλύπτεται από πλευρά Ατλαντική Συμμαχία συνέχεια που έπρεπε να είναι ευρωπαϊκή. Στη Λευκή Βίβλο βλέπετε απαντήσει από ευρωπαϊκή σκοπιά. Άρα μηνύματα ε, ε, μιας ε, διανοητικής προσέγγισης αλλαγής σε γαλλικό επίπεδο για το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Περιβάλλον υπάρχει. Είναι κάτι αξιοσημείωτο. Και ε, ζει η στρατηγική του 2020. αλλά βασίζεται επί ευαισθητοποίηση από πλευρά Ευρωπαίων πολιτών για το πρόβλημα, αλλά οι συνέπειε σε παγκόσμιο επίπεδο των απαντήσεων δεν είναι το αντίστοιχο. Είμαστε οι μόνοι που επιφορτιστήκαμε με το πρόβλημα. Και οι νέοι πόλοι δεν το κάνουν αυτό στον ίδιο βαθμό ή το κάνουν σε μια λογική βεσφαλινιακή. Συγγνώμη που το λέω έτσι απλουστευμένα. Ε, τρίτον, όσον αφορά τη ιδέα του πολυπολικού κόσμου, ε, έγραψα ομιλίες κατά το παρελθόν, εδώ και 15 χρόνια, όσον αφορά την ανάγκη να προχωρήσουμε προς πολυπολικό κόσμο. Είμαστε ρεαλιστές. Είναι διεθνής δαρβινισμός ε, ο πολυπολισμός σήμερα. Αν αυτό το λάβουμε υπόψη και λέμε ότι θα υπάρξει μια όμορφη πολυπολική κοινωνία στο μέλλον, λυπούμε, θα είναι ένας κόσμος ε, ομής βίας και σχετισμών δυνάμεων. Δεν θα πρέπει να ικανοποιούμεθα θεωρώντας ότι περνώντας από τον μονοπολισμό στον πολυπολισμό έχουμε πρόοδο. Είναι σφαλμένη και υπεραπλουστευμένη η προσέγγιση. Αυτό που είναι σημαντικό και ομολογώ ότι αυτό ίσως να φαίνεται σαν Εάν θέλουμε, πρέπει να επιθυμούμε να, να έχουμε μία ε, κατεύθυνση. Δεν είναι το πολύ που ανοίγει Πολύ δεν σημαίνει ότι ανοίγονται δύο Σημαίνει ότι ε, κάτι διασπάται, ότι χάνεται το κοινό συμφέρον. Τι, κανένα δεν διαχειρίζεται την κατάσταση, κανεί δεν έχει την, το συμφέρον, ο καθένα κινείται για τον εαυτό του. Αν θέλουμε να έχουμε πολυπολικό κόσμο και να υπάρχει ένας πλουραλισμός που είναι κάτι ε, που πρέπει να το δούμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα κοινό συμφέρον μέσα σε όλα αυτά. Ή αν μιλάμε για διαπολικό κόσμο, όπου οι σχέσεις μεταξύ πόλων θα πρέπει να καλλιεργείται, να τον επιμελούμεθα και να τον οργανώνουμε. Εκεί ναι, αλλά το σύνθημα και ο τύπος πολυπολισμός είναι η λύση ή ε, είναι καλύτερη διοργάνωση από το μονοπολικό ή διπολικό, λυπούμε, αλλά θεωρητικά εκεί υπάρχει αδυναμία, δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε τέτοιου είδους μοντέλα. Ε, δεν θέλω ε, να να βρω κάποιους τύπους και κάποιες διατυπώσεις, αλλά προσπαθώ να σας κάνω καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να λέμε λόγια και να πιστεύουμε ότι πάμε προς συνεννόηση των εθνών και μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιο. Θα ήταν ευκταίο, καλό θα ήταν κάτι τέτοιο, αλλά, ε, αλλά αντί για κονσέρτο τελικά θα είχαμε μια μεγάλη κακοφωνία και θα την πληρώσουν οι λαοί τελικά. Ήδη βλέπουμε τις συνέπειες. Τώρα συμβαίνει. Η μη διαχείριση των κρίσεων ξέρουμε τι σημαίνει σε ένα πολυπολικό κόσμο. Το βλέπουμε τα μάτια μας. Το βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Τώρα, όσον αφορά το σημείο που δεν μου, από τον κύριο Κάμπελ δεν μου απευθύνθηκε. Ο Ιαχήμ Μπίτερλιχ νομίζω ότι θα αναφερθεί σε αυτό. Δεν μου έθεσε άμεσα. Το θέμα του ΝΑΤΟ. Το θέσατε το θέμα και το ερώτημα. Βέβαια κύριε Βουλευτά, το ΝΑΤΟ, το είπα έτσι πολύ γρήγορα, στη λογική που ακολουθούμε, είναι ο απαραίτητο εταίρος μας. Αναμφισβήτητο αυτό και είναι, θα ήταν παράλογο να δούμε τα δύο αντίθετα. Διότι μόνο συμπληρωματικότητα μπορούμε να ακολουθήσουμε στη λογική μας. Το ίδιο το ΝΑΤΟ διερωτάται όμως. Ε, το ΝΑΤΟ ε, συμβιβάστηκε στην αντίληψη μεταξύ παραδοσιακή αποστολή και των νέων εξελίξεων, τη διαδρομή που θα ακολουθήσει. Και ήδη στην σύλληψη, στην αντίληψη μου ανέπτυχθε τι θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Ήμουνα στη γειτονία, πήγα στην Καμπούλ, εκεί βλέπουμε σημαντικέ αλλαγέ μετά από μια επώδυνη φάση μια αποστολή που ε, κατέληξε, ολοκληρώθηκε και δεν ολοκληρώθηκε ταυτόχρονα. Και θα πρέπει από εκεί να συναγάγουμε συμπεράσματα και μαθήματα και να μην τα επαναλάβουμε αυτό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ έγκυται η λύση. Α δούμε τα τελευταία γεγονότα, την κρίση στη Γεωργία. Εκεί τα είδαμε τα μάτια μου. Το ΝΑΤΟ δεν μπορούσε να δράσει. Και κατά κάποιο τρόπο δεν έπρεπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολήθηκε, δεσμεύτηκε ε, περισσότερο από την πολιτική σκοπιά από τη στρατιωτική Δηλαδή πριν, πίσω από τους πολίτες στείλαμε στατιωτικούς ε, μη εξοπλισμένους και ε, ήταν ένα είδος πολέμου πενταήμερου. Ε, δεν υπάρχει όμως μια λύση μοναδική και αποκλειστική. Λιβύη, ναι, εκεί μπορέσαμε να προσφύγουμε στον ΝΑΤΟ υπό ορισμένε προποθέσει σε κάποια όρια που όλοι γνωρίζουν πολύ καλά εδώ οι παριστάμενοι. Κοιτάξτε με το Μαλί, βλέπουμε τι μαθήματα παίρνουμε από εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα πρέπει να παραδεχθούμε χωρί ε, από την αρχή να προδικάζουμε τα πράγματα υπέρ Χρειαζόμαστε έναν ρεαλισμό. Α, γι' αυτό καλούμε. Θέλουμε ρεαλισμό. Και κανεί που έκανε τι παρουσιάσεις δεν, αρκείται σε λόγια και σε ε, μεγαλόσχημες δηλώσεις. Αντίθετα, θέλουμε ευαισθητοποίηση ξεκινώντας από την πραγματικότητα που είναι σαφέστατη. Τέλος. Ε, πιστεύω ότι ξεκινώντας από αυτά που έχουμε μπροστά μας, τα δεδομένα, το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο θέλουμε να ξαναρχίσουμε ποιο είναι το φάσμα των ε, ευθυνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέματα ασφάλειας και αμήνης δεν στέφεται κατά κανενός, αλλά κατά της κρίσης που αντιμετωπίζεται, της γενικευμένης κρίσης. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε, διότι επιβάλλεται από τον κόσμο σε εμά. άρα είναι ευαισθητοποίηση που ζητούμε και σίγουρα όχι επιχειρηματολογία για μια διοργάνωση ε, αντιπαράθεσης με τα μαθήματα του το Αφγανιστάν και τα όρια του ΝΑΤΟ και τα όρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως βλέποντας αυτά θα πρέπει να εργαστούμε. Ήρθε η ώρα. Ξέρουμε ότι πολιτικά δυστυχώς ε, εμπόδια εμποδίζουν τις συναλλαγές. Αλλά όταν αντιμετωπίζουμε όλοι τέτοιες προκλήσεις, είναι και η ώρα να εξετάσουμε το θέμα σοβαρά και να εργαστούμε. Και τις δικές του απαντήσεις ο κύριος Πίτερλινγκ. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε στον εκπρόσωπο των Εγγλέζων να του μιλήσω στα αγγλικά. Κοιτάξτε, για μένα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και εγώ εργάστηκα για αρκετό καιρό στην πολιτική. Ξέρω ένα πραγματικό φίλο Ευρωπαίο, το Helmut Kohl. Το ΝΑΤΟ για μας ήταν πάντα η σπονδυλική στήλη, η επιτυχημένη σπονδυλική στήλη του παρελθόντος. Μόνο που ο κόσμος γύρω μας ε, άλλαξε ριζικά το ΝΑΤΟ αναζητά αυτή τη στιγμή το μελλοντικό του ρόλο. Κυρίως λόγω του Αφγανιστάν και των εξελίξεων εκεί που για μένα δεν αποτελούν επιτυχία. Αυτή είναι η δική μου ε, στρατιωτική άποψη. Μόνο που οι Αμερικανοί φίλοι μας, ε, αυτοί θα καλέσουν εμάς τους ε, Ευρωπαίους να επιδείξουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Θα υπάρξει αλλαγή των δομών, το ΝΑΤΟ θα αναλάβει άλλα καθήκοντα. Αυτό λοιπόν για μας τους Ευρωπαίους σημαίνει ότι εμείς, ε, εμείς οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουμε διαφορετικές αποστολές, αλλά σημαίνει επίσης ότι εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει επιτέλους ε, να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στη συνεργασία, να μάθουμε ε, να χειριζόμαστε καλύτερα το θέμα το οικονομικό και πρέπει να σας πω ότι σε κάποιες ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι για τα εξοπλιστικά προγράμματα και για τους ε, διαγωνισμούς που έλαβαν χώρα. Και εγώ διαπιστώνω ότι οι ευρωπαϊκοί στρατοί υποχρηματοδοτούνται. Από το 90 με απασχολεί το θέμα που ήμουν τότε σύμβουλος ασφαλείας. Τότε το θέμα αφορούσε τη Γαλλία και σε επισκέψεις στο Βρετανικό στρατό και εκεί ενημερώθηκα για ακριβώς το ίδιο. Άρα δηλαδή πρέπει να ζητήσουμε κάποιες μορφές της εξειδίκευσης, του pooling και sharing, της συνεργασίας, να βρούμε κάποιες άλλες δομές. Τρίτον, η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ημών και μου είναι το ότι εγώ πιστεύω στους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κρίνω απολύτως απαραίτητους. Βεβαίως δεν θα μπορέσουμε εδώ να κάνουμε τη συζήτηση για το ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο αυτού, κύριε Ευρωβουλευτά. Και κατ' ουσίαν ε, μπορεί να μην δίστανται τόσο πολύ οι απόψεις μας. Μόνο που εγώ διαπιστώνω το ίδιο περίπου με εσάς, με κάποια πικρία βέβαια, με μια επίγευση πικρίας. Τα τελευταία 20 χρόνια χάσαμε πολλά, κυρίως την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην Ευρώπη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν στα τέλη φθινοπόρου του 1991 με μια γαλλογερμανική πρωτοβουλία προτείναμε την, να βελτιωθεί με αρχή τότε η γαλλογερμανική με, να εξοπλιστεί καλύτερα ε, τότε είχαν όλοι συμφωνήσει ότι πρέπει να προάγουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Γι' αυτό λοιπόν γνωρίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία όπως και τότε σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς ε, δεν υλοποιήθηκε και ανταυτής ε, πρόκειψε ένας οργανισμός ε, και πολλοί μας κατηγόρησαν ότι αυτό ήταν προδοσία στη συμμαχία και αναγκαστήκαμε να δηλώσουμε ε, τι ακριβώς ε, επιθυμούσαμε. Μόνο που διαπιστώνω ότι αυτό τότε ήταν μια απόλυτα σωστή ιδέα. Ίσως να ήταν πολύ νωρί. Ε, μπορεί, μπορεί αυτό ίσως να συμβαίνει. Όμως ήταν σωστό να διαμορφωθεί διαφορετικά η συνεργασία. Και μόλις τώρα διάβασα ένα γερμανικό έγγραφο ενός γνωστού φιλοευρωπαίου όπου προτείνεται οι γερμανικές και οι γαλλικές αεροπορικές δυνάμεις ε, να συστήσουν ε, ένα κοινό σώμα μαχητικών αεροσκαφών. Κοιτάξτε, πράγματι πρέπει να ζητήσει κανείς ε, τους τρόπους, τη δυνατότητα. Γιατί με εντυπωσιάζει και απογοτεύουμε φρικτά ε, για το μαχητικό αεροσκάφος ε, που υπάρχει στην Ευρώπη. Δύο μόνο τύποι, ένας, μια γαλλική και μια γερμανική εκδοχή. Το γαλλικό βέβαια κάλλιστα τα πάει στο Αφγανιστάν, το γερμανικό ξεχάστε το, δεν τα πάει καθόλου καλά. Άρα δηλαδή κάτι πρέπει να αλλάξει οι στόχοι που έχω κατά νου είναι, η στόχη να είναι ευρωπαϊκή. Ένα κράτος μόνος του τίποτα δεν μπορεί να καταφέρει. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους φιλοξενούμενους μας και για τον χρόνο που διέθεσαν και κυρίως για τις απαντήσεις που έδωσαν. κλείνουμε τη σημερινή συζήτησή μας με μια ανακοίνωση, πληροφόρηση. Στις 20 του Φλεβάρη, το διευρυμένο Προεδρείο της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας αποφάσισε να συντάξει γνωμοδότηση σε περίπτωση που οι επιτροπές λείπε να σας παρακαλέσω έτσι για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας και εγώ ησυχία παρακαλώ για να ολοκληρώσουμε νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε στις 20 Φεβρουαρίου το διευρυμένο Προεδρείο της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας αποφάσισε να συντάξει γνωμοδότηση σε περίπτωση που οι επιτροπές ΛΥΠΕ, ή ΙΤΡΕ αποφάσισαν να συνάξουν ψήφισμα αντί για έκθεση πρωτοβουλία για την Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Το διευρυμένο Προεδρείο της ΑΦΕΔ αποφάσισε στις 17 Ιουνίου να ορίσει τον κύριο Κέλα ως συντάκτη μερικών τροπολογιών που θα βασίζονται στην προηγούμενη του έκθεση. Οι τροπολογίε αυτέ θα σταλούν με μορφή επιστολή στην Επιτροπή ΙΠΚΟ, η οποία θα τι ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματο. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στι 8 Ιουλίου. Έχετε λάβει τι τροπολογίε αυτέ σε μορφή επιστολή. Τα μέλη των διαβριμένων Προεδρείων τη ΣΕΤΕ και τη ΑΦΕΤΕ έχουν ω αύριο 20 Ιουνίου για να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσει. Ο κύριο Κέλλαμ είναι παρόν για να ανταλλάξει απόψεις με τα μέλη της υποεπιτροπής μας επί των τροπολογιών και να ακούσει τις τυχόν παρατηρήσεις σας. Εάν έχετε επιπλέον παρατηρήσεις, μη διστάσετε να τις υποβάλλετε στους συντονιστές της πολιτικής σας ομάδας έως αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κιάλαμ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι κάπως συνήθιστη αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει όμως να προσαρμοστούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Πάντως, αντιλαμβάνομαι ότι ο στόχος της Προεδρίας και της ΑΦΕΤ και της Επιτροπής μας είναι να προσδιορίσει το ρόλο και το μήνυμά μας στο κοινό ψήφισμα το Harbor και Σβάπ. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο και από αυτή την άποψη και με αυτό το πνεύμα στηρίχθηκα στην περσινή μου έκθεση που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο. Ε, κατέθεσα μερικές τροπολογίες. Ευτυχώς δεν πρόκειται για μια φιλεγόμενη καινούργια έκθεση, δεν είναι επίμαχο το θέμα και θα ήθελα με τους συναδέλφους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της έκθεσης του Νοεμβρίου να προτείνω διεύρυνση κάποιων τομέων που είναι απαραίτητοι ώστε να λάβουμε υπόψη και τις εξωτερικές σχέσεις. Επίσης, να τονίσω ότι στην έκθεσή μου μιλώ για το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που θα πρέπει να είναι οριζόντιο θέμα σε όλες τις εξωτερικές μας σχέσεις και επίσης ε, να προστατεύσουμε και τις αποστολές μας από απειλές ε, στον κυβερνοχώρο, αντίστοιχες ε, απειλές. Κάτι άλλο που απαιτείται είναι να αναφέρουμε την εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τον κίνδυνο εξαπόλυσης επίθεσης στον κυβερνοχώρο κατά, κράτ, κατά μιας χώρας. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω και το θέμα της νοοτροπίας ε, της διαχείρισης του κινδύνου. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ε, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν κάπως συγκεχημένη στρατηγική ο μόνος τομέας είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Ήταν το μόνο σημείο στο οποίο ήταν κάπως αόριστη εκεί η Επιτροπή. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση προς τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνουν προγράμματα για την αφύπνιση, την καλύτερη συνειδητοποίηση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο και περιλαμβάνουμε και ζητούμε να συμπεριληφθούν σε σχολικά προγράμματα ε, μαθήματα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ώστε να γίνεται καλύτερη χρήση του κυβερνοχώρου. Άλλο σημαντικό θέμα της γνωμοδότησης είναι η διαχείριση μιας εδεχόμενης ε, κρίσης στον κυβερνοχώρο, στα πλαίσια της γενικής προσπάθειας ε, διαχείρισης των κρίσεων. Χαίρομαι που η Επιτροπή εμένει στην ε, συνθήκη της Βουδαπέστης και θεωρεί ότι δεν χρειάζεται νέο διεθνής νομοθεσία για το θέμα αυτό. Συμφωνώ με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απλώς καλούμε τρι... τρίτες χώρες να προσυπογράψουν τη συνθήκη της Βουδαπέστης καθώς και τις χώρες μέλη που ακόμη δεν την κύρωσαν να το κάνουν το συντομότερο δυνατό. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και αποτελεί ένα πρακτικό πρόβλημα είναι η μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την ε, εγρήγορσή τους, την ετοιμότητά τους να εκπονήσουν εθνικές στρατηγικές ε, ασφάλειας του κυβερνοχώρου. Καλό θα ήταν λοιπόν να πιέσουμε κάπως την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να τηρήσουν αυτή την υποχρέωση, αυτό το καθήκον. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. It has been calculated that more than a million... Έχει υπολογιστεί ότι κάθε μέρα έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο ε, επιθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν η καινούργια πολιτική ασφάλειας ε, που πρότεινε η κυρία Άστον αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα πολιτικό και απαραίτητο βήμα. Για τη δική μου την πολιτική ομάδα είναι πολύ σημαντικό να την χάνε γνώριση σε το ότι ε, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και ειρήνη και η κυβερνοασφάλεια ε, δεν θα πρέπει να διεισδύει στην ιδιωτική ζωή ε, να υπάρχει προστασία δεδομένων. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Φοβάμαι ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει ε, σαφής στρατηγική για το πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά στην πρακτική και φοβάμαι το ίδιο ισχύει και για το σχέδιο έκθεσης της ΙΜΚΟ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουν οι συνάδελφοί μας από τη ΛΥΜΠΕ. Και όσον αφορά τις ε, προτάσεις της Υποεπιτροπής, ε, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία ε, στην προστασία των δεδομένων και στη μεταφορά των δεδομένων αυτών σε τρίτες χώρες. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι με τις τροπολογίες, αλλά ίσως ορισμένες εξ αυτών να μην είναι απολύτως απαραίτητες. Όπως αναφέρεται στην κοινή επιστολή, τεχνολογίες αφορούν ε, τις, ε, τα θέματα ασφάλειας, αλλά κάποιες εξ αυτών ξερούνται, όπως αν τους χάνει η 9α. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς προτείνουμε να διαγραφούν. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι να παραμείνουμε στοχευμένοι στα θέματά μας για να είμαστε πιο ε, πιστευτοί. Επίσης έχω κάποιες ιδέες για την διαφορετική διατύπωση δύο-τριών Προτάσουμε, μερικούς χάνει στο 7α, ε, γίνεται λόγος για την επικείμενη συμφωνία ε, της ρήτρα αλληλεγγύης και την ανάγκη ε, να λαμβάνονται υπόψη οι κυβερνοεπιθέσεις. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και μία προστίκη από απόφαση του Συμβουλίου που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβρη η Επιτροπή και η Πατή Εκπρόσωπος ε, από το 2015 ε, θα παρουσιάζουν μια κοινή έκθεση για τους κινδύνους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτή η αξιολόγηση κινδύνου θα αφορά και τους κινδύνους που απορρέουν από κυβερνοεπιθέσεις. Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε και το ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν κοινέ ασκήσεις ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Τέλος, πρέπει να ομολογήσουμε ότι νιώθω άβολα με αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 23, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν νέα νομικά εργαλεία σε διεθνές επίπεδο. Δεν είμαι σίγουρη για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και όπως ανέφερε το ψήφισμα ή η απόφαση του κυρίου Κέλλαμ, δεν υπάρχει ακόμα ορισμός της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας. Ε, διότι η κυβερνοασφάλεια ε, μπορεί να ε, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα αυτού του θέματος. Και όσον αφορά μία αντίδραση, οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ως όπλα και κατόπιν τούτου γιατί να πρέπει να αποκλείεται η δυνατότητα του να υπάρχει ένα ειδικό διεθνές καθεστώς που θα ρυθμίζει αυτά τα εκρεμή θέματα. Σε τελική ανάλυση, αν το σκεφτούμε σοβαρά, αυτή η δήλωση είναι και σε αντίφαση με τη δήλωση της τροπολογίας 22β. Πώς μπορούμε λοιπόν να προάγουμε λύσεις σε διεθνείς οργανισμούς αποκλείοντας απριόρι την ανάγκη συμφωνιών. Εγώ λοιπόν θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν μπορούσαν να υπάρξουν διευκρινήσει σε αυτά τα θέματα και δυνατόν θα παρακαλώ να ακούσω και την άποψη της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Η... The Commissioner, ε, αν θέλουν να απαντήσουν. Κύριος Κέλλα. Καλησπέρα, εργάζομαι στη DG Connect. Είναι κοινή στρατηγική, όπως ξέρετε. Ο λόγος της δήλωσης για τη στρατηγική και την καταπολέμηση των προβλημάτων του κυβερνοχώρου είναι ότι δεν χρειαζόμαστε νέε διεθνεί συμβάσει για την κυβερνοασφάλεια. Είναι κάτι που απορρέει από τις διεθνείς συζητήσεις που συνεχίζονται. Συχνά είδαμε να ζητούνται νέες συνθήκες σε διεθνές επίπεδο για ασφάλεια. Κάτι που δικαιολογείται από θέματα λογοκρισίας, πραγματος χάρη, ε, η ρύθμιση του διαδικτύου. Όπως ξέρετε, από το διαδίκτυο πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και ελεύθερο. Λοιπόν, ε, ήταν ένα νομικό μέσο αυτή η σύμβαση που προτείνεται. Αξιολογούμε το Συμβούλιο της Ευρώπης εξετάζει την αποτελεσματικότητα με την πάροδο του χρόνου. Συζητούνται και διάφορα πρωτόκολλα για να επικαιροποιηθεί η σύμβαση. Για την ώρα δεν ζητούμε τη θέσπιση νέων μέσων, δεν βλέπουμε να υπάρχει τέτοια ανάγκη. Δεν θέλουμε να απειλήσουμε την ελευθερία του διαδικτύου. Από την άλλη πλευρά, σε διεθνέ επίπεδο υπάρχουν άλλε διαδικασίε που εστιάζονται περισσότερο επί αρχών. Όπω η πρωτοβουλία για υπεύθυνη συμπεριφορά στον κυβερνοχώρο Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τι γενικέ αρχέ που πρέπει να διέπουν τι δράσει των κυβερνήσεων και τη βιομηχανία στο διαδίκτυο. Ελευθερία τη έκφραση, προστασία ιδιωτική ζωή, κάτι που είστε προηγουμένω, ελεύθερο εμπόριο, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων κλπ. Αυτά υποστηρίζουμε τώρα ω ε, προσέγγιση σε επίπεδο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλαμ έχει να δώσει κάποια απάντηση. Uh, Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την ε, υποστήριξη καταρχήν των τροπολογιών. Όπως σας είπα, ήταν ασυνήθιστη αυτή τη φορά η διαδικασία. Να κάνω κάποια σχόλια. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι περιμένουμε έναν ε, λογικό ορισμό του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Δύσκολο να βρεθεί ένας τέτοιος ορισμός, αλλά τονίζουμε την ανάγκη να υπάρχει. Επίσης, θέλουμε κάποιους ελάχιστους κανόνες συμπεριφοράς και στους καλών πρακτικών. Και, και σε διεθνές επίπεδο αυτή είναι η πιο πρακτική προσέγγιση και ρεαλιστική. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ως προς την ανάγκη, πιθανή ανάγκη μιας νέας διεθνούς σύμβασης αλλά θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι απόψεις και των εταίρων μας, της Κίνας, της Ρωσίας. Οι χώρες αυτές αντιλαμβάνονται, αντιλαμβάνονται πολύ διαφορετικά τα θέματα αυτά. Τώρα για το 9α. Οι τροπολογίες, επαναλαμβάνω, προήλθαν από την αρχική μου έκθεση η οποία υπερψηφίστηκε. Και απευθύνω έκκληση στη δημιουργία ενός πλαισίου για αμφίδρομη ρομή πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε εμπιστοσύνη και να έχουμε πραγματική συνεργασία με τον ιδιωτικό γιατί εκεί είναι που εμφανίζονται οι περισσότερες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία σε αυτή τη σχέση ε, και ε, να είναι υποφελής και για τις δύο πλευρές. Η επόμενη μας συνεδρία είναι 10 Ιουλίου. Ευχαριστώ πολύ.